So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε. Το, το πρώτο θέμα που έχουμε σήμερα στην τη διάταξη είναι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνιακά θέματα. αρχίζουμε νέες σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία. Ο εισηγητής μας για αυτό το θέμα είναι ο Δανιέλ Κασπάρη. Οπότε του δίνω και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια που σου άρχισε στα αγγλικά, εσύ θα συνεχίσω κι εγώ στα αγγλικά, λέει ο κύριος Κασπάρη. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε σύσταση για διαπραγματεύσεις για μελλοντική συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Με μια φιλόδοξη πρόθεση να εμβαθύνουμε περισσότερο και να ενισχύσουμε περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις που έχουμε με τη χώρα αυτή. Το 2015, για παράδειγμα, τα εμπορικά αγαθά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία ήταν το ύψος 8,1 δισεκατομμύρια. Οπότε, προ, σύντομα μάλλον, θέλουμε να έχουμε και συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και το Κοινοβούλιο αποφάσισε να έχει ένα τελωνιακό πλαίσιο πιο ασφαλές και πιο φιλικό όσον αφορά τις σχέσεις των δύο πλευρών και να υπάρχει διοικητική αρρωγή σε τελωνιακά ε, ζητήματα. Και αυτό από τον Ιούλιο. Είναι ένα βήμα παραπάνω προκειμένου να βαθύνουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη 75 συμφωνίες ε, τέτοιου είδους συμφωνιών, δηλαδή αμοιβές διοικητικής συνδρομής με τον Καναδά, τον Χονγκ την, την ε, Κίνα, την Ιαπωνία. Οπότε ήρθε η στιγμή τώρα να έχει μια τέτοια συμφωνία και με τον αξιόπιστο αυτόν εταίρο μας που είναι η Νέα Ζηλανδία. Σήμερα συζητάμε για τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία αυτή είναι συμφωνία από την οποία θα υποφεληθεί το θεμητό εμπόριο, έχοντας πιο φιλικές ανταλλαγές. Θα υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία των τελωνιακών αρχών για να μπορούμε πιο εύκολα να χρησιμοποιούμε τα νέα μέσα ή να τα κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά. Θέλουμε να προωθήσουμε σύγχρονες διαδικασίες για να κερδίζουμε σε χρήμα και χρόνο, δημιουργώντας επίσης και συνεργασία υπό ίσιους όρους. Επίσης, θέλουμε να αποφύγουμε παραβάσεις των τελωνιακών κανόνων και έτσι να μην φτάνουν παράνομα αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω, συνάδελφοι, τη στήριξή σας, να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη, προκειμένου να έχουμε μια καλή και στενή συνεργασία στον τελωνιακό τομέα με τη Νέα Ζηλανδία, κάτι το οποίο θα βαθύνει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτή τη, αυτή τη γλυκή, γλυκιά συμφωνία να την υποστηρίξουμε. Ναι, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι πολύ καιρό στο Συμβούλιο και χαίρομαι που το συζητούμε. Η συμφωνία για τα τελωνιακά ζητήματα θα βοηθήσει να κάνουμε πιο ε, ισχυρή τη συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία. Αυτή η συμφωνία είναι επίσης σημάδι για μια καλύτερη συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι ένας αξιόπιστος σημαντικός ε, ε, εταίρος. Το έχουμε δει και με τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Μιλάμε για αμοιβαία συνδρομή στο τομέα των τελωνιακών ζητημάτων. Αυτό είναι μια σημαντική βάση για συνεργασία. Θέλουμε να επιτύχουμε κοινούς στόχους όπως είναι η νόμιμη ε, εμπορία προϊόντων έτσι ώστε να έχουμε προμήθεια ε, προϊόντων και ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας. Νομίζω λοιπόν ότι ε, με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο ε, τις νομικές διαδικασίες βελτιώσει, αλλά θα έχουμε και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο, κυρίως όταν μιλάμε για παραβίαση των διατάξεων. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα εγγυηθούμε και την προστασία των πολιτών, αλλά και την εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη, την αξιολόγηση των νέων διαδικασιών, ε, θα είναι Επίσης, ένα τρόπος ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα τελωνιακά ζητήματα, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα έχουμε ανταλλαγή προσωπικού, ε, προσωπικό το οποίο θα μπορέσει να ανταλλάξει εμπειρίες και να συζητήσει. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή το Κοινοβούλιο εδώ έχει μόνο δικαίωμα σύμφωνης ε, γνώμης, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να μην την δώσουμε και νομίζω ότι έτσι θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας που είναι πάρα πολύ σημαντικές και αναγκαίες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Κράκεν. Ε, καλημέρα Πρόεδρε. Ακριβώς στην ώρα μας θα μιλήσω εκ μέρους του συναδέλφου Κάμπεμαν, ο οποίος είναι ο εισηγητής για τη Νέα Ζηλανδία και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Το ECR χαιρετίζει τη συμφωνία. Η Νέα Ζηλανδία είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας ε, σε μια εποχή που γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση για την Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Είναι λοιπόν επίκαιρη αυτή η συμφωνία ε, για τα τελωνιακά που θα προστατεύσει το νόμιμο εμπόριο και θα βοηθήσει να απατάξουμε τις παραβιάσεις ε, ε, που γίνονται λόγω παράνομου εμπορίου αγαθών. Ε, είναι ένας τομέας διμερών διακανονισμών, όπως είναι ας πούμε η Συμφωνία για τα Τεχνικά Πιστοποιητικά και η Συμφωνία για τα Κτηνοτροφικά τα κτηνιατρικά, συγγνώμη, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν μια ισχυρή πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασιστεί μια πιο ισχυρή σχέση ε, και πιστεύω πιστεύω γενικά το θέμα θα το διαπραγματευτούμε εύκολα και γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, σύντομη και ακριβής, όπως πάντα. Ο κύριος Μπούχλερ για τους πράσινους. Να είμαι και ακόμα πιο σύντομος. Η συμφωνία είναι σίγουρα κάτι καλό. Θα την υποστηρίξουμε. Απλώς μια σύντομη παρατήρηση. Όταν κανείς ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία, το πρώτο που τον ε, εντυπωσιάζει, που προσέχει, είναι ε, ότι τον ρωτάνε αν, έχουν μαζί ε, αν έχει μαζί του κάτι το οποίο θα παραβιάσει τη βιολογική ασφάλεια. νομίζω ότι είναι λίγο αστείο μένα, αλλά καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο ότι εκεί σε επίπεδο ειδών φυτών υπάρχουν ιδιαίτερα είδη και δεν θέλουν τίποτα να περάσει για να μην τα καταστρέψει πλήρως. Ε, δηλαδή ε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, για όλα τα είδη τους και παρόλο που φαίνεται λίγο αστείο και πρέπει κανείς καμιά φορά να πάρει κάποια αστεία μέτρα, νομίζω ότι αυτό σε επίπεδο Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών δεν είναι τόσο εύκολα να το δώσουν έτσι. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε κάποιον άλλον που θέλει να μιλήσει. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΚΣ. Έχουμε τον κύριο Βέη. Έχετε το λόγο. Να μας δώσετε κάποια πρακτικά παραδείγματα. Ήμουνα στην Νέα Ζηλανδία με την αντιπροσωπεία Είπε ο κύριος Μπούχνερ κάποια πράγματα ήδη. Υπάρχουν κάποιες διαφορές λοιπόν μεταξύ μας, αλλά γενικά μου φαίνεται ότι το σύστημα είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Ε, πού χρειάζεται διοικητική βοήθεια. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Εγώ από την πλευρά μου είδα ότι η ικανότητα της Νέας Ζηλανδίας σε διοικητικά θέματα είναι πλήρως ανεπτυγμένη. Κύριε Κρέιπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Ισηγητά, αξιότιμοι βουλευτές, μπορώ να είμαι σύντομος, γιατί όλοι κάνετε μια καλή περίληψη και του περιεχομένου και των αναμενόμενων ωφελών από τη νέα αυτή συμφωνία με τη Ζηλανδία. Όπως είπα, τη Νέα Ζηλανδία είναι ένας καλός, αξιόπιστος εταίρος και μόνο πλεονεκτήματα θα έχουμε αν έχουμε πιο ανεπτυγμένη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Η συμφωνία αυτή έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την διμερή συνεργασία, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Νέα Ζηλανδία είναι γνωστή αξιόπιστη χώρα στη διεθνή σκηνή σε τελωνιακά θέματα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων. Το να έχουμε ένα τέτοιο εταίρο, το να αναπτύξουμε τη συνεργασία μπορεί να έχει ε, μία θετική επίδρα, επίπτωση πέρα από τη διμερή, στενή διμερή συνεργασία με τη χώρα αυτή. Τώρα, για το επίπεδο ικανότητας και δυναμικού των τελωνιακών αρχών της Νέας Ζηλανδίας, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι πολύ ικανή αρχή. Ίσως λόγω της θέσης της Νέας Ζηλανδίας, λόγω της παράδοσης της Βρετανικής που υπάρχει στη χώρα. Ο έλεγχος των υγειονομικών και φυτογειονομικών μέτρων είναι πολύ ανεπτυγμένος. Δεν αφορά μόνο τα τελωνιακά θέματα, παρότι οι τελωνιακές αρχές συνεισφέρουν φυσικά. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να συνεργαστούμε σε όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τα έσοδα, αλλά και την ασφάλεια, την καταπολέμηση της δημοκρατίας, Φερρυπίν, αλλά και την ασφάλεια των προϊόντων η ασφάλεια των προϊόντων είναι εμβληματικός φάκελος ε, των τελωνίων όλων των χωρών και η συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία ε, μπορεί να μας ωφελήσει γιατί θα υποφεληθούμε από την εμπειρία που έχει η χώρα αυτή για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Όμως ε, η φοροαποφυγή η φορολογική ε, παράδειση δεν είναι ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ή όχι. Uh, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ δεν συζητάμε φορολογικά θέματα, αλλά τελωνιακά θέματα και η φοροαποφυγή είναι θέμα άλλων συναδέλφων. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ, δεν έχω άποψη καν για αυτό το θέμα. Wäre Ενδιαφέρον. Κύριε Κασπάρη, Τάνιελ, σχόλια. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις απόψεις τους, όπως και την Κομισιόν. Θα το δούμε το θέμα στην Επιτροπή. Και αν υπάρχουν και κάποιες έτσι ελκυστικές ε, συνεισφορές από τους υπόλοιπους, θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρομαι και εγώ για την επόμενη εβδομάδα. Περνάμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα τον Ιανουάριο, δηλαδή στι ε, ε, στις αρχές του χρόνου και 20 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ για την πρώτη αυτή συζήτηση και πάμε στο σημείο 11. Ένα άλλο θέμα που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είδε σήμερα ε, μέσα στα πλαίσια της δομής των μελλοντικών ταμείων το θέμα αυτό ε, αρχίζει να λαμβάνει μεγάλη σημασία, είναι πολύ σχετικό λοιπόν. Έχουμε ε, εδώ την θέση μας που πρέπει να καταθέσουμε στην Επιτροπή Νομικών. Έχουμε επίσης την Επιτροπή Μεταφορών η οποία έχει κάποιο θέμα ε, με αυτό και ζήτησε από τους ε, συντονιστές να δώσουν μία θέση για αυτό το θέμα. Γι' αυτό δίνω στη συνάδελφο το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχετε μπροστά σας το σχέδιο της έκθεσης. Υπάρχουν έξι σημεία που θεωρεί σημαντικά ο εισηγητής. Τα έχω στα αγγλικά και θα το κάνω στα αγγλικά. Ωραία. Την περισμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο ξεκίνησε μία ε, συζήτηση για τους ίδιους πόρους, για να διευρύνουμε τον προπολογισμό της Ένωσης λόγω των μεγάλων οικονομικών προκλήσεων που υπάρχουν μπροστά μας και στο εγγύς μέλλον, αλλά και ε, πιο μακροπρόθεσμα. Το είπατε ήδη αυτό. Δεύτερον, η συνεχιζόμενη συζήτηση για τους ιδίους πόρους οδήγησε την ε, Επιτροπή Προπολογισμού να ετοιμάσει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ιδίων Πόρων, ε, επί των οποίων η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα γνωμοδοτήσει. Στο σχέδιο γνωμοδότησης, ο εισηγητής Μίλησα για γενικά θέματα, γενικού ενδιαφέροντος, αλλά ασχολήθηκα και με πιο ειδικά θέματα που αφορούν την ίντα. Γενικά, το σύστημα ιδίων πόρων και η μεταρρύθμιση του θα πρέπει να ε, οδηγήσει σε μείωση των δαπανών των ε, ε, κρατών μελών. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εθνικές συνεισφορές που βασίζεται στο ΦΠΑ και στο εθνικό ε, εγχώριο προϊόν θα πρέπει να επανεξεταστεί και η δυνατότητα για βιωσιμότητα και τελωνιακούς δασμούς που βασίζονται στις εκπομπές ε, θα πρέπει να διερευνηθεί ως μια δυνατότητα ούτω ώστε να, να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας ε, που υπάρχουν στο COB21. Επιπλέον, οι εισαγωγές ε, από ξένα προϊόντα και τα τέλη για τη ζάχαρη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αλλά θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ο προϋπολογισμός της ε, Ένωσης και επειδή μπορεί να μειωθούν αυτά τα τέλη, ε, μπορεί να μειωθούν και τα έσοδα του προϋπολογισμού. Και δεν θα πρέπει οι εθνικέ συνεισφορέ και αυτά τα τέλη να ε, τροφοδοτούν αποκλειστικά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με του συναδέλφου ε, τη Επιτροπή, ούτω ώστε να υπάρχει πλατιά συνένεση ε, σε δύο εβδομάδε που θα συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στο σκιώδη συγγετή, ο κύριος Σούστερ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει ως τώρα. Θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κοινή θέση σε πάρα πολλά σημεία. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που χρειάζεται και είναι τρεις οι λόγοι. Οι οικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν όλο και περισσότερα δαπάνε ε, που καταλογίζονται στον προπολογισμό και πρέπει να αντισταθμιστούν με έσοδα. Αυτό πρέπει να συνδεθεί στενά με την πολιτική εμπορίου, τα, γιατί έχουμε και τα διάφορα επενδυτικά ταμεία για την Αφρική που συζητούνται τώρα και άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Επίσης με το Brexit η βάση των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί δραματικά. Αυτό είναι μια οικονομική και πολιτική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει ε, ε, να περιμένουμε τουλάχιστον ότι αν έχουμε μια επιτυχημένη εμπορική πολιτική ε, θα έχουμε και αντίστοιχα ε, αυξημένα έσοδα, άρα σταδιακά να μειώσουμε και τους δασμούς. Επίσης, ε, να έρθω τώρα στο θέμα τη ε, ομάδας εμπεριογνωμόνων, οι οποίοι μιλάνε για νέα ίδια ε, για νέους ίδιους πόρους ε, που θα περάσουν μέσα από την ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες. Είναι η προστιθέμενη αρχή, αξία του εμπορίου, αλλά και η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε ίδιους πόρους οι οποίοι θα προέλθουν από φορολογικά έσοδα, για παράδειγμα, και καλύτερο συντονισμό. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θέσω, το οποίο πηγαίνει λίγο ε, πέρα από αυτό που είπε ήδη η συγγήτρια, είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση ε, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια συμφωνία για ολόκληρο αυτό το σύστημα γιατί ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις βελτίωσης που είχαν γίνει και στο παρελθόν για το σύστημα των τελωνιακών δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την φοροαποφυγή και τα και πρέπει αυτά να εφαρμοστούν πλήρως. Όπως είπα, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πολύ καλή θέση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπούχνερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς ε, συμφωνούμε με τα βασικά σημεία αυτής, αυτού του σχεδίου. Ε, μόνο μια λεπτομέρεια στο σημείο 4 λέει ότι στους τελωνιακούς δασμούς και στις εισφορές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα και οι εκπομπές. Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε ένα σύστημα που είχαμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το σύστημα πιστοποίησης για το διοξίδιο του άνθρακα αυτό μπορούμε να το συμπληρώσουμε με κάποιες, κάποια άλλα αντίστοιχα συστήματα που αφορούν τις εκπομπές όσον αφορά στην εισαγωγή ενέργειας. 400 δις ευρώ δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς ε, για την ενέργεια και αν ε, το δει καλή, κανείς αυτό προσεκτικά θα καταλάβει ότι ε, καταστρέφουμε το κλίμα μας. Στις ε, ε, λεπτομέρειες λοιπόν δεν συμφωνώ με τον εισηγητή. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να το ενσωματώσουμε αυτό στα ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θέλουμε, να, θέλουμε να είμαστε πιο στοχευμένοι, εκεί που πρέπει να υπάρχουν βελτιώσεις να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το λόγο η Κομισιό. Λουκάντα Κάραλη από τη Γενική Διεύθυνση Τρέιντ. Να πω και εγώ για το σημείο 4. Ε, εδώ και καιρό συζητούμε το θέμα των ε, πιθανών εκπομπών ε, και των πιθανού φόρου στις εκπομπές, μιλάμε για το εμπόριο των εκπομπών, Ποιες είναι οι δυνατότητες που βλέπετε εσείς μέσα στα πλαίσια ε, των κανόνων του ΠΟΕ. Ποιο είναι το περιθώριο που έχουμε για, τους χειρισμού, για χειρισμούς. Μπορείτε λίγο να μας τα πείτε πιο συγκεκριμένα. Γιατί είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή για να παίξουμε με αυτό το θέμα. Και για το σημείο 6, γιατί ο μέσα εμπορικής άμυνας, ε, δεν είναι μια σταθερή ε, πηγή πόρων, αλλά είναι πηγή πόρων. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσο μεγάλη πόσο μεγάλη έκταση έχουν αυτοί οι δύο πόροι, αν υπάρχουν διακυμάνσεις κτλ. Ε, αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και εκεί αναφέρονται ζητήματα σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα Οπότε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Με ε, πιέζετε ουσιαστικά να μπω στις λεπτομέρειες για το σημείο 4. Όντως είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα πώς δηλαδή θα προχωρήσουμε και με το φόρο άνθρακα. Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα διαθετηθεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων και θα έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα εσωτερικό σύστημα ε, φορολόγησης του άνθρακα ανάλογα με το αποτύπωμα άνθρακα. Για το σημερινό σύστημα, το εμπορίου δηλαδή δικαιωμάτων, δεν είναι φτιαγμένο σαν ένα σύστημα συλλογής φόρων. Παίρνει κανείς ε, δωρεάν δικαιώματα εφόσον ξοκάχονται από κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με την παραγωγή. Υπάρχουν προκλήσεις δηλαδή για το πώς θα μπορέσουμε αντίστοιχα να καταλήξουμε σε κάποιο φόρο στα σύνορα, ανάλογα δηλαδή με το αποτύπωμα άνθρακα. Δεν είναι σαφές ε, λοιπόν αν έχουμε ένα φόρο που θέλουμε να θεωρήσουμε κάτι σαν ισοδύναμο με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων στα σύνορα, πώς θα γίνει αυτή η ισοδυναμία. Γίνεται η συζήτηση σε θεωρητικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε ανάλογα με το πώς παράγεται ένα προϊόν, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικά παραδείγματα στην ομοθεσία μας. Υπάρχει οδηγία για τις ανανόσιμες πηγές ε, ενέργειας που έχει διαφορετικά κριτήρια βιωσιμότητας καυσίμων και συγχρόνως έχουμε και ένα σύστημα για να καταγράψει το αποτύπωμα άνθρακα των διαφόρων ε, προϊόντων μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής, με την ενέργεια που χρησιμοποιείται κλπ. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα. Είναι κάποιες πρώτες διακρίσεις που θα μπορούσαμε εδώ να σας δώσουμε και από εκεί και πέρα το εξετάζει και από αυτό. Τώρα για το δεύτερο θέμα, για τα μέσα εμπορική άμυνα, δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, αλλά στην απόφαση λέει ότι όλα τα έσοδα που απορρέουν από αυτό γίνονται ε, παντός είδου δασμοί δηλαδή, οι έσοδα γίνονται ήδη πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντύπωσή μου είναι πάντως ότι όντως πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό, ένα 2% των εισαγωγών. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος των ιδίων πόρων από τους τολωνιακούς δασμούς. Αλλά πρόκειται για κάτι αρκετά σταθερό τον τελευταίο καιρό. Οι τελωνιακοί δεσμοί συνολικά, έτσι, 15 με 20% των ιδιοπόρων. Πολύ λιγότερο βέβαια από το ΦΠΑ και από το GNI, το εθνικό εισόδημα. Πρόεδρος, ωραία, έχουμε τριμερή διάλογο για τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους ίδιους. Έχετε μια ερώτηση, παρακαλώ. Να πω ότι αυτό το εργαλείο δεν φέρνει ε, έσοδα, οπότε δεν χρειάζεται καν να ανταλλάσσουμε και προϊόντα. Ναι, λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα. Το Μάιο περιμένουμε να έχουμε πρόταση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και κάποιες ιδέες για τους ίδιους πόρους, σωστά. Ναι. Αυτή είναι η γραμμή για την Άνοιξη. Αλλά πρόσφατα δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, Γοντελίβε, θέλεις εσύ να απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ του εισηγητή σε όλο το θέμα βλέπω δύο τεχνικά ε, ζητήματα. πώς ε, θα διατυπώσει η Κομισιόν την πρότασή της για τους ίδιους πόρους. Για μας ε, όμως πολιτικά είναι πιο σημαντικό το ψυχολογικό ζήτημα. Εμπιστεύεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσωποποιείται στην Κομισιόν ώστε να υπάρχει ένα τελικά σόφρον σύστημα για τους ίδιους πόρους το οποίο θα το καταρτήσει αυτή ή θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Ε, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Και κάτι άλλο, η Κομισιόν για άλλη μια φορά προσπαθεί να ε, τελειοποιήσει την ε, στρατηγική, την επικοινωνιακή της για να μην μπορεί καλή να την ανατρέψει. Ευχαριστώ. Ναι, και η πολιτική εφαρμογή των ιδίων πόρων θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα και στα κράτη-μέλη πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Ίσως να υπάρχει ε, δυνατότητα να έχουμε ε, με την ε, προστασία από τις καταστροφές και την προστασία των συνόρων μια σύνδεση μεταξύ των δαπανών, δηλαδή σε αυτούς τους τομείς, με τα έσοδα. Αυτά θα τα δούμε όμως. ευχαριστώ η προθεσμία για τροπολογίες είναι η επόμενη εβδομάδα 27 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα και μετά θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο την έκθεση. 22, 23. Ωραία, ευχαριστώ. Ήμασταν γρήγοροι. θα μπορούσαμε να ε, κάνουμε ένα άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι πιο κάτω, η παρακολούθηση. Δεν ξέρω ακριβώς αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος που πρέπει να είναι εδώ. Δεν είναι εδώ οι άλλοι συγκεκριμένοι. άρα θα έχουμε ένα διάλειμμα 20 λεπτά.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Okay, so... Ωραία, πριν ξεκινήσουμε, μία ανακοίνωση. Ο κύριος Μόιζερ έφυγε από την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών και τώρα είναι μη εγγραμμένο μέλος. Άρα οι σοσιαλιστές και δημοκράτες σήμερα έχουν μόλις 9 μέλη και όχι 10. Ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Πριν όμως γίνει αυτό, ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Για να βάλετε λοιπόν την κάρτα σας, αρχίζει η ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. I mean, And close the Κλείνω τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν ε, τις ψηφοφορίες μας με το σημείο 12 προς μία στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. Μαριέτε Σάκε είναι η συγκήτρια. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία να πω ότι η κυρία Πικίνα συνυπέγραψε 22 τροπολογίες της κυρίας Ρέντινγκ. Είναι στην ψηφοφορία, στο έγγραφο των ψηφοφοριών, αλλά όχι στις τροπολογίες. Άρα, πολλές από τις τροπολογίες συμπίπτουν. Αυτά είχα να πω. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 66 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη από την ε, τροπολογία 97. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και άλλη προσθήκη, η 96 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. 96 άρχεται η ψηφοφορία. And Πέρας. Απορρίφθηκε. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος, 106, προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε. 130 λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ, πέρα της προφορίας, εγκρίθηκε. Οι επόμενες καταπίπτουν και πάμε στην τροπολογία 135 και 136 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 137 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Ήρεμα, ήρεμα, εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Α, όχι. Πρέπει να πάμε πίσω, να ψηφίσουμε την 141. Υπέρ παρακαλώ, της 141. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα πάμε στην 142, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα της 142. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 152. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 153. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκατόν πενήντα οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία του ΕΛΚ για την έγκριση της σύστασης του Κοινοβουλίου υπέρ της τροπολογίας αυτής κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την προφορική αυτή τροπολογία στην 158 που λέει σύμφωνα με τις συστάσεις που έδινε το Κοινοβούλιο. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Να σηκώνετε καλά τα χέρια σας παρακαλώ. 159 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε 159, οπότε δεν πρέπει να ψηφίσουμε την 161. Ωραία. 159 λοιπόν πάλι. Ποιοι είναι υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 159. Ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Όντως εγκρίθηκε. Να σηκώνετε καλά τα χέρια. Για τελειώσει. Είναι περίπλοκο, δεν μπορώ να σας δω. Μετά βλέπω μόνο τα κατά και λέω ότι απορρίφθηκε, ενώ δεν είχα τις τα χέρια στα υπέρ. 160 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 162, υπέρ. Αποχές, λέει ο πρόεδρος. Ναι, κατά ήθελα να πω. 162. Ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 184. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. 185 υπέρ,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 Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβατική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28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 Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 45. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε 46. Όχι. 47 διορθώνει ο πρόεδρος. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά 47. Ψηφίστε. Τέλος και εγκρίθηκε. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα των σοσιαλιστών υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. Την προφορική τροπολογία στην 8 τη συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την αιτιολογική σκέψη. Έτσι. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίθηκε. Μάλιστα. Πάμε στις νομοθετήσεις ανά επιτροπή. Επιτροπή Ήτρε καταρχήν. Προσοχή εδώ. Έχουμε μία τροπολογία της Ήτρε. Ε, που υιοθετήθηκε γιατί ψήφισα μια άλλη τροπολογία. Πάμε στην Ήτρε 4 υπέρ. Κατά. Πάλι δεν είναι σαφές. Ξανά τα χέρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ήτρε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι υιοθετείτε αλλά το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την Ήτρε 8. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Ήτρε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η Ήτρε 13. Καταπίπτει. Η Ήτρε 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν γιατί υιοθετήσαμε τις αντίστοιχες τροπολογίες. Πάμε στην ΙΜΚΟ. ΙΜΚΟ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την ΙΜΚΟ 1. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα ακόμα ηλεκτρονικά. Πέρας χωρίας Απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 3 καταπίπτει. ΙΜΚΟ 5. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ήμκο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. Ήμκο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ήμκο 14. Καταπίπτει. και η 15. Πάμε στη 17. Ήμκο 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πάμε τώρα στη Λίμπε. Λίμπε 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Λίμπε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Λίμπε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Λίμπε 6 υπέρ. Κατά. Εποχές Υιοθετείτε. Λίμπε 8 υπέρ. Ξανά παρακαλώ τα χέρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Λίμπε 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την Λίμπε 13. Πέραση της ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Υιοθετείτε. Λίμπε 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα συνολικά την έκθεση την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Το ΕΛΚ έχει έναν βουλευτή παραπάνω. Πέρας φοφορίας. Ευρεία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Υιοθετείτε με πλατιά-πλατιά πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στη Μάριέτε Σάκε. So, now we are... Και τώρα πάμε στο επόμενο μεγάλο φάκελο. η αναθεώρηση για τη διπλή χρήση. Εκατόν πέντε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμό 8 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Το προφορική τροπολογία της Μαρή Βεστάγκη υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, άποχες, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 13. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφέστατα απορρίπτεται. Και τώρα. 123 και 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 και 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας το ελέγξω όμως ηλεκτρονικά. 125 και 126. Πέρας φοφορίας απορρίπτεται. Συμβασμός 8α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 152, Είναι προφορική τροπολογία που αντικαθιστά την παλιά. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155 και 156 πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές υιοθετούνται. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, άποχες. Ας το τσεκάρουμε το 100, την 162 εκτονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας απορρίπτεται. 22. Τοπολογία 22 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τρεις α, ίδιες τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετούνται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 12 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 192 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 13 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 14 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Προφορική τροπολογία του Κρίστοφερ Φιέλνερ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 208. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας, υιοθετείτε. 209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 210 υπέρ, κατά, άποχες την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τη 210. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 216. Υπέρ. Ναι, είναι μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι την, την ψηφίσαμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 216. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε φωνικά την 218. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σε δύο τμήματα τώρα. Τη 221. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι δεν είμαι σίγουρος. Ε, ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος. Το δεύτερο, του δεύτερου τμήματος 221. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Διαθετείτε. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Διοθετείτε. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 15 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός 16 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 243 και άφετ 24 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετούνται. 207 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 248 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 249 υπέρ κατά αποχές. Δεν είμαι σίγουρος. Ελέγχουμε εκτονικά την 249. Πέρας προφορίας απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε χρονικά. 253. Πέρας προφορίες. Υιοθετείτε. Εξακαλύπτει και 254 και 255. Και πάμε στην 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. Του, 257 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 258 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι υιοθετείται αλλά την ελέγχουμε χρονικά. Πέρας. Υιοθετείται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά την ελέγχουμε. 262 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. 39. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά 263. Πέρας φοβορίας. Υιοθετείτε. Α. Καλά το είδατε. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 39. Ένα εξωφορίας. Πέρας. Υιοθετείτε. 266 υπέρ. Κατά. Εποχές. Μάλιστα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 266. υπέρ φοφορίας. Υιοθετείται. Συμβιβασμός 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 294 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται συμβασμός 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβασμός 19 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 20 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Άφετ τροπολογία 32 της άφετ δηλαδή υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 310 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Άφετ. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 318 και 34 υπέρ. Ξέχασα την 317. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 318 και 34 απνάφετε Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 319 και άφε 35 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 320 υπέρ. Κατά. εποχέ. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές. Τι ψηφίζουν. Υπέρ. Ελέγχουμε 320. Ηλεκτρονικά. Ε. Υιοθετείτε. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 20α. Περ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 323 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 324 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 21 υπέρ. Κατά. Εποχές Υιοθετείτε. Πιθανή προσθήκη στην τροπολογία στην 21 είναι η 326 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται 328 και 329 υπέρ κατά εποχές τις ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτονται. 330 και 331. Όχι μόνο την 330. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Άφετ. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 335. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 340 και 341. Υπέρ κατά εποχές υιοθετείται 343 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται συμβασμός 23 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε. Προλογία 37 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 348 υπέρ Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά το, την, την 348. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 2α υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 69 υπέρ κατά, κατά αποχές σας παρακαλώ ακόμα μια φορά την 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 3 υπέρ. Όχι πίπτη, συγγνώμη. Η τροπολογία 3 όχι της ΑΦΕΤ αλλά του εισηγητή. Τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 76, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Είχαμε ψηφίσει και την 77 και την 78 για το, την αιτιολογική σκέψη 11, βέβαια, όλες μαζί. Έτσι. Όχι υπέρ. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Μετά συμβιβασμό 3α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Έχουμε μία ψηφοφορία on block 152. Υιοθετήθηκε ήδη. Είστε σίγουρος. Γραμματεία. Πάμε στην τροπολογία 6 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5. Ξάφετ. Περ. Κατά. Αποχές. Δεθετείτε. Συμβασμός 4. Υπέρ. Α, όχι. Πρώτα την 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Μετά, μετά τρεις πανομοιότυπες τροπολογίες. 89, και τις υπόλοιπες υπέρ, κατά, αποχές υιοθετούνται. Τροπολογία 7 της άφετ, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 8 της άφετ, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Δύο ίδιες τροπολογίες, υπέρ, κατά, αποχές. Τις ελέγχουμε. Την 92 δηλαδή και την 9 της άφετ. Έναρξη προφορίας. Πέρας. Υιοθετείτε. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 6. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 30 υπέρ κατά όχι, όχι, είναι αιτιολογική σκέψη 30 και έκανα λάθος. Τροπολογία 12 φυσικά. Περ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 100. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 103 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας υιοθετείται. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Και τώρα πάμε στο δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Ένα S&D. Εγκρίνεται, όπως σας είπα. 358 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 351. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 352. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. 300. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι και αυτή απορρίπτεται, αλλά να τη ελέγξουμε. 353 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 354 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 355 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 356 υπέρ. Κατά.

Εγκρίνεται λοιπόν 335, άρα καταπίπτουν αυτέ οι τροπολογίε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο 367. 367 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 371 υπέρ, κατά, άποχες, απο, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 374 υπέρ κατά άποχες να ελέγξουμε. 374. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 375 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. 376 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 377 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 380 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 381 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 381. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 384 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 386 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 387 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. 387. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is... Hmm. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 388 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 389 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 390 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 395 υπέρ κατά απορρίπτεται 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 396 υπέρ Συγγνώμη, 398 διορθώνει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται. 400 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 402 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 55 υπέρ αποχές απορρίπτεται 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 407 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 408 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 409 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Α, αυτό ε, κατέπιπτε. Άρα 410 από τον Κρίστοφερ Φέλνερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλδημοκράτες τίποτα. 410. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλλον είναι υπέρ, ε, φαντάζομαι. πέρας της ψηφοφορίας. Και όντως εγκρίνεται. 57 υπέρ. ακαταπίπτει Άρα, 411. 411 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Άρα η επόμενη καταπίπτει και μετά πάμε στην 415 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 419 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία 419 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 424 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε όπως τροποποιήθηκε την έκθεση άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. Με μεγάλη, πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια στον Κλάους Μπούχνερ και στην διαπραγματευτική ομάδα. Τώρα δίνω το λόγο στον εισηγητή. Θα ήθελα ε, ε, να έχω εντολή για άμεση ε, ε, διαλλαγή και συνομιλία με το Συμβούλιο. Να το ψηφίσουμε λίγο και αυτό. Άρα, να ξεκινήσει άμεσα ο τριμερής διάλογος. Αυτό είναι ε, που ψηφίζουμε υπέρ. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Θα πάμε στην Ολομέλεια λοιπόν και περιμένω μετά από τη συζήτηση και την ψηφοφορία για τις τροπολογίες να πάρουμε την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων στον τριμερή διάλογο. Ωραία. Συνεχίζουμε και περνάμε στο σημείο 14. Είναι της Αντιπροέδρου Σάιφη, πρόκειται για την ατήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Έχουμε πρώτα τη συμβαστική 7. Υπέρ,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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, συμβαστική 4 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και 26 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 26. Μπορείτε να ψηφίσετε. Εγκρίθηκε. Τροποποιημένη έκθεση τώρα. Παρακαλώ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Σάιφη. Και περνάμε στην τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα. Πρόκειται για προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κρυμαία και την Σεβαστούπολη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας τη ψηφοφορία. εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία ψηφοφορία που είχαμε. Και τώρα, όποιος θέλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει ησύχως παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε παραπέρα στο 16, την έκθεση για την παρακολούθηση των ομάδων. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Επιτροπής μας. Είχαμε στις 12 Οκτωβρίου μια τέτοια παρακολούθηση για τις σχέσεις με τα Ηνωμένε Πολιτείες με τον Διευθυντή και τον πρώην διαπραγματευτή Γκαρσία Περσέρο, Ιγνάσο Γκαρσία Περσέρο και τον Τζον Κλάρκ από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη που ήταν και αυτός εκεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα που έχουμε, όπως είναι οι ελιές, το κρέας, ε, ζητήματα σχετικά με τη γεωργία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ. Δεν φαίνεται τελικά σε ποια κατεύθυνση θα πάνε, τα, ε, θα πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, που θέλουν να καταλήξουν και επίσης ε, δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης ε, για την εθνική ασφάλεια, ειδικά το άρθρο 2 και το 3.2, καθώς ο Τραμπ έχει δραστηριοποιηθεί στο θέμα της ε, βιομηχανίας Χάλιβα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν Φλεβάρι-Γενάρη. Επίσης, ε, πριν από την ε, Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπένος Άιρες θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε από κοινού να προσπαθήσουμε να μην υπάρξει πάυση αυτών των διαπραγματεύσεων ειδικά στην διαδικασία έφεσης για τους ε, ε, δικαστές, δηλαδή να μην ε, μπλοκάρεται το εφετείο περαιτέρω. Άρα, κυρίως οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι σε αυτό το πλαίσιο. Μετά στις 17 Οκτωβρίου έγινε μια ομάδα παρακολούθησης για την Ιαπωνία με τον βασικό διαπραγματευτή Μάρο Πετιτσιόνα. Μας μίλησε για την ε, κατάσταση και φαίνεται ξεκάθαρο ότι η συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη. Ε, αν και η Επίτροπος εχθές μίλησε για κάποια ανοιχτά ζητήματα. Στις 18 Οκτωβρίου είχαμε την ομάδα για την ε, Νότια Ασία, ειδικά μίλησαμε για το Πακιστάν και το GSP+. Καρίμ, μπορείς να μας κάνεις μια αναλυτική παρουσίαση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, έλαβε χώρα αυτή η Επιτροπή με εκπροσώπους από το Πακιστάν στις 23 εδώ στις Βρυξέλλες, στο Κοινοβούλιο. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Μάλεκ και Φαντουργίας και τον Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Σαφαλή. Οι συνομιλητές μας συνοδεύονταν και από τον υπεύθυνο εμπορίου στην ε, πρεσβεία του Πακιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους, όπως επίσης από το Κοινοβούλιο του Πακιστάν. Η συνάντηση αυτή εδώ στις Βρυξέλλες έγινε ακριβώς πριν από τις συζητήσεις που γίνονται αυτή την ε, εποχή για την ε, εφαρμογή της συμφωνίας GSP-SYN. Ε, θα μας παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκθεση στις αρχές, το πρώτο τρίμηνο του 2018 και θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν τότε να συζητήσουμε την ε, θέση μας. Όσον αφορά τώρα το Πακιστάν, όσον αφορά την αξία των εισαγωγών βάσει του GSP-SYN, Μιλάμε για 70% εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη συμφωνία αυτή, το καθεστώς δηλαδή τη συμφωνια αυτης αυτή GSP-SYN. Έχει υπάρξει πρόοδος από το Πακιστάν όσον αφορά την νομοθετική πρόοδο ε, επίπεδο δικαιωμάτων, σε θεσμικό μάλλον επίπεδο. Παραμένουν όμως διάφορες προκλήσεις όσον αφορά τη θανατική ποινή, τα δικαιώματα των παιδιών, τους βασανισμούς και θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμμόρφωση ε, στον νόμο, ε, διαφθορά, ε, θέματα κυρώσεων λόγω βλασφημίας, ελευθερία έκφραση κλπ. Τώρα, ο υπουργό ε, που ήταν παρόν στη συνάντηση είπε ότι η συμφωνία GSP συν δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο, έχει να κάνει και με την τήρηση υποχρεώσεων, με αποτελέσματα δηλαδή υπέρ του ΛΟΤΟ του Πακιστάν. Τονίστηκε επίση ότι πρέπει από τη δικιά μας ε, την πλευρά να κοιτάξουμε τι θα γίνει και μετά το 2023. Η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να είναι το τέλος των φιλοδοξιών μας. Ο Υπουργός ε, ξέφρασε την πεποίθησή του ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνε χέρι-χέρι και υπάρχει πρόοδος. Τώρα για τις δυσκολίες. Αναφέρθηκαν ομοσπονδιακές δυσκολίες όσον αφορά το σεβασμό των μηχανισμών που υπάρχουν τώρα σε επίπεδο επαρχιών. Οπότε υπάρχουν μέτρα για τις διάφορες επαρχίες, κυρίως μετά την ε, υλοποίηση της GSP συν, αλλά τώρα πρέπει να ενισχυθεί και ο ομοσπονδιακός χαρακτήρας. Πάντως υπάρχει πρόοδος. Σημειώνουμε επίσης ότι δεν φτάνει μόνο η έγκριση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά είναι θέμα εφαρμογής, πώς θα περάσουν όλα αυτά στην πράξη και πώς θα υπάρξει διαφοροποίηση εξαγωγών. Μέχρι τώρα βασίζονται κυρίως στην υφαντουργία και σε έτοιμα ενδύματα, στο έτοιμο ενδύμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση και βελτίωση της σχέσης business to business και ε, σχέσεις μεταξύ πακιστανικών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών. Εμείς ευχαριστήσαμε όλους τους συναδέρφους βέβαια που συμμετείχαν με τους αξιωματούχους τους στη συνάντηση αυτή και τονίσαμε ότι η ενισχυμένη συνεργασία με την συμφωνία GSP-SYN είναι κάτι που απαιτεί και την επίσκεψη ειδικών απεσταλμένων από διεθνείς εμπορικούς οργανισμούς. Ε, το Πακιστάν είπε ότι ευχαρίστως. Συνολικά ήταν μια καλή ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να ανταλλάξουν απόψεις προκειμένου να ετοιμαστούν για την αρχή της επόμενης χρονιάς που θα υπάρχει σχετική έκθεση της Κομισιόν που θα μας ε, παρουσιαστεί. Τώρα, όσον αφορά την ε, Νότια Ασία γενικώ, θα ήθελα να πω κάτι για τη Σρι Δεν θα πάρει πολύ. Ο λόγος που θέλω να το κάνω αυτό είναι ότι ανησυχώ και περισσότερο για την ε, κατεύθυνση του ταξιδιού. Πολύ πρόσφατα επαναφέραμε την ε, Σρι στο σχέδιο αυτό για μια GSP συν και το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού προσπάθησε να μας ε, καθησυχάσει για την μελλοντική κατεύθυνση. Συναντήθηκα όμως με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρα Πάρνα, εδώ στις Βρυξέλλες και δυστυχώς φαίνεται ότι η συνάντηση ήταν μάλλον καταστροφική. Γιατί έκανε πίσω σε δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργό με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι ισχύουν τα όσα είχαμε πει από την αρχή. Αλλά χτες μόλις έμαθα άσχημα νέα από τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σρι Φαίνεται ότι όντως υπάρχει οπισθοχώρηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν απέναντί μας. Οπότε ελέγχουμε την κατάσταση. Ίσως όμως να ζητήσω επιγόντως να επανέλθει το θέμα ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος έγκαιρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρύμ και ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε για τη Σρι Λάνκα. Γνωρίζετε ότι ετοιμαζόμαστε για τη Σριλάνκα, οπότε καλό θα ήταν να γνωρίζουμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ωραία. Τώρα έχουμε και το Μερκοσούρ, 19 Οκτωβρίου. Εχθές ε, μιλήσαμε στην Επιτροπή διεξοδικά για το θέμα. Στις 7 Νοεμβρίου υπήρξε η ομάδα για την Ασία. Ο Ντέιβιτ Μάρτιν θα μας κάνει την παρουσίαση γι' αυτό. Ευχαριστώ. Στι 17 Νοεμβρίου κάναμε μια συνάντηση για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή συναντηθήκαμε για να εστιάσουμε για την στην Ιντονισία, όπου είχαμε μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν. Αλλά αυτά που μα είπαν ήταν απογοητευτικά για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Στο τελευταίο γύρο έγινε στι 11 έω 15 Σεπτεμβρίου στι Βρυξέλλες ε, από ό,τι φαίνεται οι Ινδονήσοι ε, οπισθοχωρούν ε, στις δεσμεύσεις τους σε σχέση με τα όσα είχαμε στο κείμενο. Ε, στο κείμενο. Ας πούμε στα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά έχουμε πιστοχώρηση. Οι Ινδονήσοι ε, δεν δέχονται τη δεσμεύσή τους να διαπραγματευτούν την πρόσβαση στην αγορά για τις δημόσιες ε, συμβάσεις. Πρόοδος για τις επενδύσεις στα αγαθά και τις υπηρεσίες είναι αργή και στο δικό του σύστημα οι Ινδονήσοι λένε ότι πρέπει να κάνουν εσωτερική διαβούλευση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το συζητάνε μαζί μα, ούτε καν. Θετικό ποιο είναι, το εξή. Ένα. Στο IPR, δηλαδή δικαιώματα ε, πνευματική ε, ιδιοκτησία, εκεί δέχονται GNI, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, θετική ε, εξέλιξη. Επίσης, ε, ε, ετοιμάζουν μία ε, διαπραγμάτευση ελευθερών εμπορίου με την Αυστραλία. Άρα είναι αλλού το μυαλό τους, αλλού η εστίασή τους. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, στη δική μας FTA, στη δική μας Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου δεν υπάρχει πρόοδος. Το θετικό είναι ότι μας είπαν ότι μέχρι το 2018 μάλλον θα κλείσει αυτή η ιστορία. Από ό,τι μας είπε όμως η Κομισιόν αυτό είναι υπεραισιόδοξο να τελειώσει δηλαδή, το θέμα μέσα στο 2018. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ για το Brexit έχουμε την ομάδα παρακολούθησης. Θα ήθελα να συζητήσουμε τις διαβουλεύσεις του ΠΟΕ για τις ποσοστώσεις και τους δασμούς και την προσαρμογή τους. Φυσικώς, το θέλαμε αυτό να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι δυστυχώς η Κομισιόν απέρριψε την πρόσκλησή μας. Κάνουμε πολλές διαθεσμικές συζητήσεις για το θέμα αυτό και τελικά θα κάνω μια συζήτηση στην Επιτροπή Άρα, τελειώσαμε εδώ με το σημείο 16 και το 17 είναι η συνάντηση Καριφόρμ. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Καριφόρμ. Ο Ντέιβιτ θα μας κάνει μια σύντομη ε, ε παρουσίαση για την εμπειρία αυτή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Πριν μπω όμως στο ψητό για αυτή τη συνάντηση, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους να υπενθυμίσω ότι η αντιπροσωπεία υπάρχει λόγω της Επιτροπής μας. Όταν ε, περάσαμε την ε, Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος της ε, εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Και εγώ ήμουν εισηγητής για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την Καριφόρ. Μία κοινοβουλευτική επιτροπή εξέταση όμως δεν έκανε όπως έπρεπε τη δουλειά της. Είναι μόνο η τρίτη φορά που θα συνεδριάσει τώρα αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Κάναμε δύο στο 2013, μέσα στο 2013 και για τέσσερα χρόνια τίποτα. Το καλό είναι όμως ε, είναι ότι συναντηθήκαμε τελικά και ότι κάναμε μια ειλικρινή, όπως λέει η διόγλωσσά μας, ας πούμε, συζήτηση, που στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστή, πολύ καυτή. Η πλευρά της ε, Καριφόρν δεν πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πολλά για να τους βοηθήσει οικονομικά κυρίως και να, τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ΕΠΑ, της, οικονομικής... Ε, της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Εμείς είπαμε ότι τα διάφορα τα κονδύλια που τους δίνουμε ε, τα υποδαπανούν. Και δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη μία θέλουν περισσότερους πόρους και από την άλλη. Ας πούμε, έχουμε μια πραγματικότητα όπως το Επενδυτικό Ταμείο για την Καρεβική, ε, το Ταμείο Βοήθεια για το Εμπόριο, ε, όλα αυτά τα ταμεία στα οποία έχουν δικαίωμα να εκταμιεύσουν ποσά, ε, εκεί υπάρχει υποχρησιμοποίηση. Εάν θέλει περισσότερα κονδύλια, πρέπει να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί αυτά που έχει ήδη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι παρά το γεγονό ότι δεν συναντηθήκαμε για τέσσερα χρόνια, πολλά από τα θέματα ξανάρχονται, επανέρχονται κτλ. Είναι τα θέματα που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Ένα εσωτερικό θέμα το οποίο μας ενοχλεί είναι τα λιμενικά τέλη που αφορά τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη. Και θεωρούν ότι είναι μια στρέβλωση ανταγωνισμού. Θεωρούν ότι τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη έχουν πλεονέκτημα που αυτοί δεν το έχουν. Οι υπόλοιπε δηλαδή, τα υπόλοιπα εδάφη τη Καραϊβική. Και του επίση πολλά από τα κράτη τη Καραϊβική είτε λόγω έλλειψη πολιτική βούληση ή λόγω έλλειψη διοικητικού δυναμικού που τελικά είναι το ένα ή το άλλο, μάλλον και τα δύο είναι, εξαρτάται από τη χώρα δεν έχουν εφαρμόσει την μείωση των ε, δασμών ε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε συμφωνήσει ή λόγω πολλών περιπτώσεων έλλειψης, ε, σε πολλές περιπτώσεις είχαμε έλλειψη δημο, διοικητικού δυναμικού για να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Αυτό είναι, που είναι σίγουρο είναι ότι δεν έχει γίνει η σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση. Όμω το 2015 υπήρχε ένα νέο σχέδιο δράση, ούτω ώστε να δώσει μια νέα ορμή στην Συμφωνία και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδο στι γεωργικέ ενδείξει ε, για τη γεωργία, στα πολιτιστικά προϊόντα, στα, ε, στη Συμφωνία Αμοιβαία Αναγνώριση και τη Ε, άρα υπάρχει έτσι κάποια κίνηση. Ένα από τα σημαντικά πράγματα για του, τα νησιά τη Καρυβική είναι το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Γιατί εμείς ε, θέλουμε να προστατεύσουμε τις δικές μας γεωγραφικές ενδείξεις, κυρίως εμείς δηλαδή. Αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν ε, προϊόντα, ας πούμε, σε συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο τομέα, ας πούμε, και να τα προστατεύσουν. Ε, έχουν να κάνουν αυτά με το τσάι και άλλα προϊόντα. πήγαμε σε μία εγκατάσταση κοκοφινίκων Ε, έρευνας για το κακάο, υψηλής ποιότητας, ε, με σπόρους και τα λοιπά και ποικιλίε. Και το κακάο του Τρινιδάδ ε, πουλιέται στο Χάροντζ. Οχτώ με δέκα φορές σε, ψηλότερη τιμή από την κλασική ας πούμε, τιμή του κακάου. Θέλουν δηλαδή να ε, χωθούν σε αυτή την ειδική αγορά, ας πούμε. Ε, γενικά όμως, ούτε η παρακολούθηση ήταν καλή της ε, συμφωνίας, ούτε η πρόοδος, ούτε η, πρόοδος, ούτε παρακολούθηση λοιπόν. Τώρα όμως υπάρχει ευτυχώς πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές για να λειτουργήσει και αυτό είναι το θετικό. Ναι, πέρασε καιρός και θα έπρεπε να έχουμε ε, καλό αποτέλεσμα, αλλά το δουλεύουμε. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Όχι, ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. David. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Γιατί ελπίζω ότι σε δύο λεπτάκια ο Επίτροπος Μοσχοβησί θα έρθει. να συζητήσει τις εξωτερικές μας σχέσεις και τη μακροοικονομική τους διάσταση. Δύο λεπτά διάλειμμα. Okay, let's Περνάμε στο σημείο 18 και πολύ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Μοσκοβισή και έτσι έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε να μας μιλήσει για τις εξωτερικές οικονομικές μας σχέσεις Υπάρχει πρόταση για εμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Υπάρχει και η εξωτερική διάσταση των τελωνίων. Και βεβαίως στην Επιτροπή μας έχουμε και την μακροοικονομική αρρωγή προς κάποιες χώρες με τις οποίες έχουμε, τις οποίες έχουμε εταίρους. Οπότε έχουμε πολλά κοινά στις αρμοδιότητές μας, κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι, ε, Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και σήμερα το πρωί παίρνω το λόγο στην Επιτροπή σας. Είναι η πρώτη μας συνάντηση και σας ευχαριστώ θερμά που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση. Όντως υπάρχει μια διεθνής διάσταση στα οικονομικά, είτε πρόκειται για τα φορολογικά, τα χρηματοπιστωτικά, το διεθνές εμπόριο Και γι' αυτό, επειδή είμαι υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα, με ενδιαφέρει η Επιτροπή σα, τα τελωνία, γιατί πρόκειται για τα εμπορεύματά μας ε, που μπαίνουν και βγαίνουν από τα σύνορά μας, οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση του διεθνούς εμπορίου. Υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας βέβαια και η σχέση της ασφάλειας με το εμπόριο. Έχω και τα τελωνιακά στην, ε, στις μου, στο χαρτοφυλάκιό μου που επίσης έχουν και εξωτερική διάσταση. Βγαίνω από μια τέτοια συνάντηση όσον αφορά την μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων. Πολύ θα ήθελα ε, λοιπόν να σας πω ότι στις 5 Δεκεμβρίου θα συζητηθούν και θα ήθελα να ακούσω και από εσά για να δούμε σε τι κυρώσεις τελικά αποτρεπτικές θα καταλήξουμε. Είδατε ποιες είναι οι προβλέψεις του φθινοπόρου για τις τάσεις στο εμπόριο. Επιταχύθηκε η οικονομική δραστηριότητα τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο εξάμεινο σε σχέση με τα 7 τελευταία χρόνια. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να δούμε τι γίνεται στις ε, αναδυόμενες χώρες, στην Κίνα για παράδειγμα, που υπάρχει τεράστια οικονομική ανάπτυξη Στη Ρωσία και τη Βραζιλία επίσης ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, οπότε γενικά οι χώρες BRICS συμπεριφέρονται καλύτερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Και γενικά η διεθνής οικονομική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί στα πλαίσια του 8% και το 2018 και 2019 περιμένουμε 4%. Η ευρωπαϊκή που είναι 2,3% είναι η πιο μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Είχαμε δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτή η ανάπτυξη ευρωπαϊκή θα πρέπει να στηριχθεί και στην ε, παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι το 2019 θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και στις αναδυόμενες χώρες. Η συναλλαγές εμπορικές θα αυξηθούν πάνω από 4% το 2018 και 2019, περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει την Άνοιξη. Αυτή λοιπόν είναι περίπου η κατάσταση, το πλαίσιο της, ε, το οικονομικό. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα συζητάμε για τη διεθνή ε, διάσταση των τελωνιακών. Είχαμε 300 300 νούμε εκατομμύρια δηλώσεις που συλλέχτηκαν στα σύνορα και εξετάστηκαν. Καταλαβαίνετε ότι είναι και θέμα ασφάλειας των εξωτερικών μας σύνορων. Εμείς συμμετέχουμε σε μια διεθνή αλυσίδα παραγωγής που γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Γι' αυτό και πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να εντοπίζουμε τις απάτες και άρα χρειάζονται οι πιο αποτελεσματικοί δυνατόν έλεγχοι. Είτε από το 2014 έχουμε πει ότι πρέπει να ε, ενταθεί η συνεργασία μας η διμερής με όλους τους εμπορικούς μας εταίρους για να αντιμετωπιστεί η απάτη, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για να εντοπίζουμε τους κινδύνους καλύτερα και η συνεργασία μας αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ε, πολυμερές πλαίσιο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων. Έτσι όπως έχει σήμερα η κατάσταση, τα τελωνία ενδιαφέρουν ακόμα περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, γιατί συνεισφέρουν επίσης και στην προστασία μας από τη διεθνή τρομοκρατία. Διότι κόβει τα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα είτε ονομάζεται Daesh, το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, καταφέρει να πουλήσει στην ευρωπαϊκή αγορά ε, αρχαία, τα οποία βέβαια παράνομα βάζει μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό και έκανε πρώτα κανονισμού επιτροπή πρόσφατα, μιλώντας για την εισαγωγή αυτή αρχαιοτήτων, και οι τελωνιακές αρχές τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή αγορά από τέτοια εμπορεύματα. Περί τίνος πρόκειται. Όσοι εισάγουν ευαίσθητα τέτοια προϊόντα θα πρέπει να έχουν κάποια άδεια. Είτε πρόκειται για ε, αρχαία, είτε πρόκειται για έγγραφα παλιά, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία άδεια. Θα πρέπει να φαίνεται ότι εξάγονται νόμιμα τα αντικείμενα αυτά. Θα υπάρχει επίσης και η λασιμότητα με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε την αγορά μας, να προστατεύσουμε και αυτά τα αρχαία. Συνεπώς η πρόταση αυτή ε, συνοδεύεται από μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης αλλά και από την κατάρτιση των τελωνιακών με τη βοήθεια και της UNESCO. Πρέπει να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο δηλαδή τελωνιακοί μας με αυτήν τη διάσταση. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός γενικότερου σχεδίου αντιμετώπισης της τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, έχουμε ενημερώσει τους κανόνες για τον έλεγχο των εισόδων και εξόδων ρευστού, ε, το ίδιο και με τα ταχυδρομεία. Έχουμε μιλήσει επίσης για τις ε, χρεωστικές κάρτες, τις προπληρωμένες μάλλον, και για τα πολύτιμα μέταλλα. Όλα αυτά είναι προτάσεις που πολύ σύντομα θα καταλήξουν. Επίσης και για την αντιμετώπιση των απατών στο ΦΠΑ. Γιατί και αυτό είναι κάτι που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Μιλάμε για πάνω από 50 εκατομμύρια το χρόνο. Γι' αυτό και θέλουμε μια καλή αντιμετώπιση των ε, απατών αυτών, των απειλών αυτών για πάτες στον ΦΠΑ. Γιατί είναι ένα ε, διασυνοριακό ζήτημα. Τώρα όσον αφορά την εξωτερική διάσταση του χαρτοφυλακίου μου για τα φορολογικά. Έχουμε τα Paradise Papers. Διαπιστώνουμε ότι κοινικά ε, χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το πλανήτη φορολογικά κόλπα για να μην πληρώνει κανείς ε, φορολογία. Είναι πράγμα που συζητιέται και στο Διεθνές Μεσονοτικό Ταμείο και στο ΝΟΣΑ και παντού για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα. Η φορολογική παράδειση πρέπει να είναι γνωστή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και εγώ αυτό θέλω. Θέλω διαφάνεια, να γίνονται γνωστά αυτά. Να υπάρξει λοιπόν ένας ευρωπαϊκός κατάλογος φορολογικών παραδείσων. Στο ΕΚΟΦΗΝ της 5ης Δεκεμβρίου θέλω να εγκριθεί αυτό. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Και οι χώρες που θα είναι σε αυτό το κατάλογο θα κληθούν να παρετηθούν από τέτοιες πρακτικές. Το θέμα δεν είναι τόσο οι κυρώσεις που θα τους επιβληθούν, όσο το να πιστούν να εγκαταλείψουν αυτές τις πρακτικές οι χώρες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο είναι απάτες που μπορεί να έχουν να κάνουν με σκάφη, με αεροπλάνα, με ιδιωτικά δηλαδή jet. Τα είδαμε αυτά με τα Paradise Papers. Οπότε στο τέλος του μήνα αυτού θα ήθελα μέτρα ώστε να βοηθήσουμε τις ε, υπηρεσίες τις κατάλληλες των διαφόρων χωρών να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Τώρα αναφερθήκατε και στη μακροοικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γειτόνες χώρες η βοήθεια αυτή έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ακριβώ επειδή υπάρχει και μακροοικονομική αστάθεια. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, το γνωρίζετε αυτό το μέσο. Στόχο του είναι η μακροοικονομική σταθερότητα και η δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών που βοηθάμε, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Πρόκειται για ένα έκτακτο μέσο, οπότε οι προτάσει επιτροπή θα πρέπει από του νομοθέτε να εγκρίνονται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είχαμε την μακροοικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Θα συναντηθώ με τον Υπουργό Οικονομικών της Ουκρανίας σήμερα το απόγευμα. Ξαναβερθήκαν πριν από μερικέ εβδομάδε. Υπάρχουν και θεσμικά βέβαια ζητήματα. Δεν μπορώ να πω και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανταποκριθήκατε στην έκκλησή μας και πάρα πολύ γρήγορα εγκρίθηκε η βοήθεια αυτή η οποία συνεισφέρει στη σταθερότητα της οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Και χαίρομαι που αναγνωρίζετε η αξία του μέσου αυτού στην γενικότερη πολιτική μας, μάλιστα τώρα που συζητάμε και στα μέσα του δρόμου το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ λοιπόν για την ε, βοήθειά σας που ήταν από 0,5 δις σε 5 ε, τον τελευταίο καιρό. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και μετά το 2020. Το πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας, η μακροδημοσιονομική μας βοήθεια στην Ιορδανία, την Τινησία, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μολδαβία που θα υπογράψουν σε λίγες μέρες οι Μολδαβοί πιέζουμε έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει και τα όσα ε, επιθύμησαν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και υπάρχει και η πρόσφατη πρόταση για μακροοικονομική βοήθεια στη Γεωργία. Συζητήσατε χθε για αυτήν και σας ευχαριστώ. Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα θα εγκριθεί και αυτή η συμφωνία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μπαίνουν προϋποθέσεις βέβαια, έτσι. Το υπενθυμίζω πάντα. Είναι η μόχλευση που χρησιμοποιούμε. Τα συζητάμε με τους ε, υπουργούς γιατί ε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες ε, κινδυνεύουν να κρατήσουν για αρκετό καιρό. Γι' αυτό και εμείς πιέζουμε και βάζουμε προϋπόθεση να γίνουν αλλαγές στις χώρες που βοηθάμε. Σας υπόσχομαι ότι η μακροοικονομική σταθερότητα και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων είναι κάτι που θα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για μας. Τώρα, τι επόμενε εβδομάδε θα δούμε κατά πόσο η Ουκρανία εφαρμόσει το υπόλοιπο πρόγραμμα για να πάρει και το τελευταίο κομμάτι της μακροοικονομικής βοήθειας. Ελπίζω. Και για τη Μολδαβία θα ε, δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο ε, τηρεί το πρωτόκολλο Μολδαβία ή όχι. Αυτά λοιπόν. Βλέπετε ότι και στον οικονομικό τομέα και στα τελωνία και στη φορολογία έχω πολλά ζητήματα στην ημερήσια διαταξή μου. Αλλά και με το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο και τους G20 και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο ε, συζητάμε πάντα. Έχουν να κάνουν τα δικά μου θέματα με αυτά της Επιτροπής σας. Πάντως θέλω εδώ να επιμείνω σε η πρόταση για τα πολιτιστικά αγαθά να εγκριθεί γρήγορα. Έχω περάσει από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και γνωρίζω ότι χρειάζονται κάποιες θεσμικέ διευκρινήσεις από την Επιτροπή. Και εγώ ήμουν εδώ ευρωβουλευτής ε, για κάμποσα χρόνια. Δεν θα σας πω εγώ ποια θα είναι η λύση που πρέπει να βρείτε. Απλώς λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια λύση αποτελεσματική. Γιατί η τρομοκρατία δεν περιμένει, συνεχίζει να χτυπάει κάθε μέρα. Οπότε, αν πιστεύετε ότι η πρόταση είναι καλή, και αυτή την αίσθηση είχα μέχρι τώρα από όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες των πολιτικών ομάδων όλων των πλευρών κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Περνάμε στις ερωτήσεις από τους βουλευτέ. Από το ΕΛΚΑ. Ο κ. Βαλέσα. Εκπροσωπώ το συντονιστή του ΕΛΚ που δεν μπορούσε να παραστεί. Έχω και μία ερώτηση ως ε, μόνιμος εισηγητής για την Ουκρανία. Ας ξεκινήσω από τις ερωτήσεις του εισηγητή, του συντονιστή. Η Κομισιόν πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ε, κακής χρήσης των ελευθέρων ε, λιμένων ή ζωνών. Και τι γίνεται με την ε, διαφάνεια, ποιος κρύβει τι και πού. Σε ό,τι αφορά τους, ε, τα paradise papers ή οποιαδήποτε άλλα papers. Είναι σωστό ότι η Κομισιόν δουλεύει για αυτό το μαύρο κατάλογο των φορολογικών παραδείσων και τον ετοιμάζει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο εργαζόσαστε και τα επόμενα βήματα. Συμπεριλαμβάνουν και τρίτες χώρες και, γιατί να, και Γιατί να μην βάλετε και τους ε, φορολογικούς παραδείσους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχέδια για την ε, παγκόσμια διανομή των φόρων, των φορολογικών εσόδων. Τώρα, για τη μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, παρακαλώ, μια ερώτηση. Στη συνάντησή μας τον περασμένο μήνα, κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για εμπορικά θέματα, καθώς και τη μακροοικονομική βοήθεια τα μέλη του ελληνικτικού Συνεδρίου για την Ουκρανία έθεσαν ένα συγκεκριμένο θέμα. Ε, η απόφαση του δεύτερου πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου και η προκαταβολική ε, εκταμίευση της πρώτης δόσης δικαιολογείται. Υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για την δεύτερη εκταμίευση της επόμενης δόσης. Της δόσης. Πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις για να εκταμιευθεί η δεύτερη δόση. Οι τελευταίες δύο δόσεις ε, αναβλήθηκαν και τελικά τον Απρίλιο του 2017 έγινε η εκταμείευση, παρότι κάποιες προϋποθέσεις δεν πληρούνταν. Σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο το πώς θα εξασφαλίσουμε την ισορροπία. Από τη μία να δώσουμε μακροοικονομική βοήθεια και από την άλλη να τηρήσουμε την αρχή της ρεσιμότητας. Ευχαριστώ. Και τώρα από το... η Αλέσια Μόσκα από τους α, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, Επίτροπε, στην Επιτροπή μας. Τα δύο πρώτα σχόλια θα ακούσετε και θα σας κάνω και ερωτήσεις. Καταρχάς, η φορολογική παράδειση. Εμεί δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ στην Επιτροπή μα με του φορολογικού παραδείσου, αλλά η ομάδα μου όμω ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Και επομένω θέλω να σα πω ότι σα υποστηρίζουμε για να συνεχίσετε προ αυτήν την κατεύθυνση. Για τη μακροοικονομική βοήθεια, και αυτό είναι για μα, την ομάδα μου δηλαδή, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Υποστηρίζουμε ότι αυτό πρέπει να είναι ένα εργαλείο που θα το χρησιμοποιούμε σωστά και είναι μεγάλη σημασία. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε το συντομότερο δυνατόν όλη τη φάση της ε, εφαρμογής και παρακολούθησης. Ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέπεια το συντομότερο δυνατόν ανάμεσα σε όλες τις σχετικές πολιτικές. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταστήσουμε αυτά τα εργαλεία αποτελεσματικά, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αυτά ήταν τα σχόλια. Τώρα, οι ερωτήσεις. Τα cultural goods, ε, τα πολιτιστικά αγαθά. Πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί αμελητή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να επιλύσουμε όλα τα εσωτερικά θέματα. Και θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις σχετικά με τις ε, σχετικές προτάσεις που κάνετε. Αν είναι αλήθεια, όπως μάθαμε, ότι το 80 90% αυτών των αγαθών, των πολιτιστικών αγαθών, ε, μπαίνουν στο εμπόριο με παράνομο τρόπο, τότε χρειαζόμαστε εργαλεία πολύ αποτελεσματικά για να υπάρχει εχνηλασιμότητα. Διερωτώμεθα, αν πέρα από την ομολογία, νομοθεσία, μέτρα και ρυθμίσεις, τι άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να πάρουμε, ούτω ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εσείς μιλήσατε για την ευαισθητοποίηση. Σωστό. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε μια σειρά από συντονισμένες δράσεις. Δεύτερον. Για να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, πώς μπορούμε οι παράνομοι εισαγωγεί να μην χρησιμοποιήσουν διάφορε κερκόπορτε για να παρακάμψουν την νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη, ένα πολιτιστικό αγαθό χαρακτηρίζεται ως τέτοιο εάν είναι ας πούμε ένα αντικείμενο 200 ή 250 χρόνων. Πώς θα κάνουμε την ηχνηλάτηση ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν άλλοι τρόποι παράκαμψης ε, της νομοθεσίας. Το θέμα είναι δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Ο κ. Σταμπάτη από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μας είπατε ότι το παγκόσμιο εμπόριο είναι μια επαρκής πηγή εσόδων και πλούτου για όλο τον κόσμο. Όμως, αυτό προκύπτει και από την ανταγωνιστικότητα της κάθε χώρας. Ας πούμε, η ισοτιμία είναι ένα πρόβλημα. Ε, μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ανταγωνιστικότητα μιας ε, χώρας. Τώρα, ας πούμε, ε, το ευρώ, η ισοτιμία του μας έχει βοηθήσει να έχουμε την ευημερία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Μιλάω τώρα για το εξωτερικό εμπόριο. Ο, το ισοζύγιο πληρωμών από το 2000 και μετά είχαμε 37 ε, δις ευρώ, ε, όταν ξεκίνησε δηλαδή η ΟΝΕ. Ναι. Τώρα έχουμε 216 δις ε, πλεόνασμα στην Γερμανία. Στην ε, Γαλλία το ανάποδο. 17 δις ευρώ ήταν το πλεόνασμα το 2000, το 2016 έλλειμμα 20 δις ευρώ. Έχει αυξήσει λοιπόν η Γερμανία το ποσοστό της στο παγκόσμιο εμπόριο από το 8% στο 9% ενώ της Γαλλίας μειώθηκε κατά το 1 τρίτο. Αυτό φυσικά έχει επιπτώσει στην εσωτερική στον εσωτερικό πλούτο της χώρας. Θα σας δώσω νούμερο. Στην Γερμανία η ανεργία τα τελευταία 10 χρόνια είναι από το 8,5 πήγε στο 4% στο 4,2% ενώ στη Γαλλία από το 8% στο 10,1%. Στους νέους η ανεργία στη χώρα σας είναι από το, 7, από το 2007 στο 2016 πήγε από το 19,5% στο 24%. Ενώ στη Γερμανία το 2007 ήταν 11,8% και τώρα έχει φτάσει στο 7,8%. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια ανακατανομή η οποία έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα της κάθε χώρας. Έχουμε λοιπόν ε, ε, νομισματική ένωση και θα ήθελα να ε, ρωτήσω την Κομισιόν. Τι γίνεται με τις διαφορετικές ισοτιμίες και τη διαφορετικά ισοζύγια της κάθε χώρας τι γίνεται με την ανάπτυξη, την εσωτερική και εξωτερική της κάθε χώρας. Παρακαλώ να τα λάβετε υπόψη σας. Και πραγματικά, κύριε Επίτροπε, θα ήμουν ευγόμενο να τα λέγατε και στους συναδέλφους σας αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους. Για την ΚΟΕ, ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που ήρθε εδώ. Ας πούμε, ε, να πούμε τώρα για την Επιτροπή για τα Panama Papers, η οποία έχει προτείνει κάποιες παραγράφους, οι οποίες θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες. Ας πούμε, οι μελλοντικέ εμπορικές ε, συμφωνίες και συμφωνίες εταιρική σχέσης ή αναθεώρηση των υφισταμένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια δεσμευτική ρήτρα για το φόρο ε, που θα συμμορφώνεται με τα στάνταρ του ΟΑΣΑ ε, και τις ε, συστάσεις ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Επίσης, οι επενδύσεις και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις μελλοντικέ συμφωνίες εταιρική σχέσης θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της θετικής στάσης. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά και τις παρατηρήσεις που κάνατε για την τρέχουσα κατάσταση ως προς τις σχέσεις μας με την Μολδαβία και την Ουκρανία ειδικότερα, αλλά ίσως να είναι και άλλες χώρες ε, που θα μπορούσαμε να πάρουμε ως σημείο αναφοράς. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση προς την Επιτροπή Εμπορίου. Πώς να το αντιμετωπίσουμε, γιατί εχθές είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για τη Μερκοσούρ και στη Συμφωνία Μερκοσούρ δεν υπάρχει μια τέτοια δεσμευτική ρήτρα. Δεν το διαπραγματευόμαστε καν και μετά έχουμε το πρόβλημα οι περισσότερες ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που έχουμε διαπραγματευτεί και ας πούμε ήδη έχουν λήξει, έχουν οριστικοποιηθεί, να μην έχουν μέσα αυτά τα στοιχεία για τη φορολογία. Τι μάθαμε λοιπόν με τις έρευνες για τα Panama Papers και τα λοιπά. Μάθαμε και το είπε και η Κομισιόν Δημοσίως ότι πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν ε, κάποια κάποιες επιπτώσεις, κάποια συμπεράσματα. Δεν πρέπει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε αυτά, αυτές τις διατάξεις στις μελλοντικές ή τις υφιστάμενες συμφωνίες. Και τώρα με τη Μολδαβία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια χρημάτων που εξαφανίζονται κάπου. Δεν ξέρει καν ο πρόεδρος της χώρας που έχουν πάει τα χρήματα, όπως λέει γενικά χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων για σκοπούς οι οποίοι είναι αμφίβολοι. Δεν μπορούμε να τους τεκμηριώσουμε, να τους ελέγξουμε κτλ. Και εφόσον έχω χρόνο κύριε Πρόεδρε, άλλη μια παρατήρηση. Δεν νομίζετε ότι ένα μορατόριο σε μια τέτοια διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών θα ήταν απαραίτητο αν δεν μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις διατάξεις. Πώς ε, ε, συνεργάζεστε με την Επίτροπο Μάλστρομ σε αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Χάουτελα για τους πρασίνους. Ευχαριστώ Επίτροπε για το θέμα των ε, συμφωνιών ε, ελευθερών συναλλαγών και τα φορολογικά ζητήματα. Να σας πω ότι όταν ο Τζόζεφ Στίγκλες πήγε στην Επιτροπή την Εξεταστική για τα Πάνομα Papers, είπε ότι θα ήταν πολύ καλό να έχουμε ρήτρε ε, για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή στις συμφωνίες αυτές, όπως μόλις μας εξήγησε και ο συνάδελφος Σόλτς. Χρειάστηκε να το συνειδητοποιήσουμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες αυτό. Επίσης, για την πρόσβαση σε τελωνιακές πληροφορίες. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα. Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις της Επιτροπής μας για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, για παράδειγμα, που ζητούν για συνολική πρόσβαση στα δεδομένα των τελωνίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αυτοποιήσουμε και να εχνηλατήσουμε τα προϊόντα που προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν ερωτήματα ως προς την βιωσιμότητα και την ηθική. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολο γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτές οι πληροφορίες σε βάση του κανονισμού των τελωνίων βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Όμως νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί πραγματικά θα αποτελούσε ισχυρό εργαλείο για τη διαφάνεια. Το έχετε τονίσει κι εσείς ως στόχο σας. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το ψηφιακό εμπόριο. Η έκθεση ΣΑΚΕ μόλις τώρα εγκρίθηκε και υπάρχουν νέες ανησυχίες που εγείρονται για την φορολογία. Πόσο μάλλον ε, για τον ΦΠΑ και την ε, αποφυγή καταβολής φόρου όταν έχουμε ψηφιακό εμπόριο. Τα εξετάζετε αυτά. Και η τελευταία μου ερώτηση για την Ουκρανία. Ποιο είναι το βασικό σας μήνυμα στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή όσον αφορά το αίτημά τους για μακροοικονομική βοήθεια. Όπως ακούμε από τις ε, παρεμβάσεις, υπάρχουν πολλές ανησυχίες εδώ στο σώμα για την έλλειψη αιρεσιμότητας ή γενικά την χαλαρή εφαρμογή της αιρεσιμότητας στις μακροοικονομικές ε, παρεμβάσεις. Ε, κύριος η ευθυντή, κύριε Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε. Τρεις-τέσσερις απλές ερωτήσεις έχω. Η πρώτη απορρέει από αυτά που είπα και ο συνάδελφος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε ένα κοινό φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αν ναι, πότε πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει. Έπειτα, θα θέλετε επίσης έναν ενιαίο συντελεστή για το φόρο εισοδήματος. Και αν ναι, τότε πότε. Και πολύ σύντομα θέλω να πω, να ο καθηγητής Σταρμπάτη εντυπωσίασε όπως πάντα με τα στατιστικά δεδομένα. Αλλά πρέπει να πω ότι η δικιά μου εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενικά στα θεσμικά όργανα και κάποιοι συνάδελφοι μάλιστα ακόμα, δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους που υποφέρουν από την φτώχεια και τη μιζέρια εξαιτία του ευρώ. Αυτό που τους ενδιαφέρει να συνεχίζουμε με όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση και να προχωράμε όλο και περισσότερο με το ευρώ. Κάνω λάθος. Ότι είναι αυτός σκοπός δηλαδή. Ή μήπως αυτά τα οποία υποψιάζομαι ισχύουν. Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο που ήρθε. Και ευχαριστώ και για το εξαίρετο έργο του όσον αφορά το, χαρτί, το φυλάκιό του και που καταπολεμάει τους φορολογικούς παραδείσους. Πολύ σύντομα θέλω να θίξω τρία ζητήματα. Πρώτον, τελωνία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δασμολογική ένωση, αλλά δεν έχει τελωνιακή ένωση. Το λέω αυτό γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου και τα λοιπά δεν είναι σαν να πρόκειται για μια τελωνιακή ένωση. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, για την εναρμόνιση ίσως θα μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά και πιστεύω ότι είναι βασικό για να στηρίξουμε και την ε, Ευρώπη απέναντι στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν ε, ε, εκείνοι που εισάγουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που τελικά περνάνε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να περνάνε εξαιτία των λοιπόν ελέγχων που έχουμε. Δεύτερον, στα θέματα συνεργασίας και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και τι ρόλο μπορεί να παίξει η δικιά μας Επιτροπή για τις ε, εμπορικές συμφωνίες. Πώ πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ώστε η συνεργασία αυτή να γίνει πραγματικότητα. Και τέλος, λαμβάνοντα υπόψη το σενάριο που έχουμε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και τις συνέπειε από το Brexit, είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει απώλεια εσόδων και άρα πρέπει να προσέξουμε τι θα κάνουμε με τις δαπάνες, γιατί αν δεν την καταστήσουμε αυτά τα έσοδα με κάτι άλλο, δεν θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Η ομάδα μας λοιπόν πάντα πίστευε ότι πρέπει να υπάρχει ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μπορείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε πώς έχει η κατάσταση από αυτού και τι θα ήταν εφικτό προκειμένου να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα έσοδά μας, γιατί τελικά οι τράπεζε είναι οι μόνες οι οποίες δεν φορολογούνται ουσιαστικά. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, λέει ο Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ωραία. Παρακαλώ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα ήθελα μια σύντομη απάντηση να δώσω, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή. Θα... Θέλω να κάνω μια ερώτηση για την Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα, αλλιώς ε, τα χάνουν. Τι γίνεται, ε, πρέπει να γίνει μια τέτοια εκταμίευση. Είναι δυνατόν να γίνει, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες τώρα όπως και στο παρελθόν. Ε, πώς ε, θα συμπεριφερθεί η Κομισιόν ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Μανουέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μοσκοβισή που ήρθε εδώ Θέλω να αντιδράσω στην ε, δήλωση του συναντέλφου από την ECR. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι συγκρίσεις που διαφωτίζουν υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα είναι και μεμονωμένες και ε, δεν είναι αμερόληπτες. Το να συγκρίνουμε, ας πούμε, τη Γαλλία με τη Γερμανία και τα βασικά οικονομικά μεγέθη, αν θέλουμε να το κάνουμε, ε, χρειαζόμαστε χρόνο για να το κάνουμε σοβαρά. Τρεις μικρές ερωτήσεις. Υπάρχει μια σχέση αναμφίβολη ανάμεσα στην οικονομική ρόμη μιας χώρας και στην εμπορική πολιτική. Η εμπορική πολιτική ε, συνοδεύεται από μια ε, σχεδόν απουσία πολιτικής ε, συναλλαγματικής. Πολλοί συνάδελφοι επέμεναν και είναι προτεραιότητα των σοσιαλιστών αυτή η ιδέα της φορολογικής ρεσιμότητας. Σήμερα έχουμε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που είναι φορολογικά τυφλές δηλαδή. Δεν θέτουν καθόλου αυτό το ερώτημα. Ενώ, τη Ενώ υπάρχουν σχετικά προβλήματα. Παναμάς. Ο Παναμάς σήμερα είναι σε μια συμφωνία ελευθέρων ανταλλαγών Κεντρικής Αμερικής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθαρός ε, δικαιούχος. Αν υπήρχε αυτή η ρήτρα ερεσιμότητας, φορολογικής ερεσιμότητας που τη θέλουμε εμείς, ίσως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεύτερο παράδειγμα για το μέλλον, έτσι, το Brexit. Σήμερα υπάρχει μια διαδικασία. Στη δεύτερη φάση του Brexit θα μπούμε, θα μπούμε μάλλον στη δεύτερη φάση στο, σε λίγους μήνες. Και προς το παρόν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυνοντές του, ε, χρησιμοποιούν ένα φορολογικό laissez-faire ε, στα στα υπερπόντια βρετανικά εδάφη και ορισμένοι θεωρούν θα γίνουν και φορολογική παράδειση. Είναι αλήθεια. Αυτή η άγουσα έχει επιλεγεί. Τότε θα πρέπει να βάλουμε, με συγχωρείτε, και τη φορολογική αιρεσιμότητα απέναντι σε αυτό τον αυριανό, ας πούμε, εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είναι ε, πολύ δεσμευτική, να έχει τα BEPS του, ΟΣ, του ΟΣΑ, τις διάφορες συστάσεις και να υπάρχει και μια επαλήθευση σύν το χρόνο, ούτως ώστε να παίρνουμε μέτρα μέχρι και την απώλεια των εμπορικών πλεονεκτημάτων ε, για αυτό που δεν ε, σέβεται. Τώρα, εγώ ήμουν ε, εισηγητής για το IMF, για την δηλαδή, μακροοικονομική βοήθεια με την Ιορδανία, προς την Ιορδανία. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να έχουν νόημα. Αλλά σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο συχνά δυσκολεύονται οι εταίροι μα. Βλέπω, α πούμε, του Ιορδανού να απαντήσουν και να ανταποκριθούν εγκαίρω στι απαιτήσει που είναι τεχνική και διοικητική φύσεω. Υπάρχουν πολλέ καθυστερήσει από πλευρά του. Και διαρωτώ με, μήπω η Κομισιόν θα μπορούσε να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποιες ε, ερωτήσεις, Επίτροπε. Υπάρχουν τελείως διαφορετικές πρακτικές των τελωνιακών αρχών, ειδικά στα λιμάνια. Υπάρχουν κάποιοι μυστικοί κατάλογοι που, για τους εισαγωγείς. Ε, τις ξέρουν αυτές και λένε αν εισάγεις το τάδι αγαθό ας πούμε θα πας στον Βούργο. αν εισάγεις κάποιο β αγαθό θα πας αλλού. Τώρα για τα πολιτιστικά αγαθά. Υπάρχουν διαφορετικές επίσης πρακτικές στις τελωνιακές αρχές απέναντι στα πολιτιστικά αγαθά. Ποια είναι η λύση, πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη σας. Επίτροπος, πολλές ερωτήσεις άκουσα. Καλωσορίζω τη δέσμευση που αναλαμβάνετε όλοι σας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, για μια ανοιχτή οικονομία, για το εμπόριο, για την ασφάλεια μέσω των τελωνίων και της ενθάρρυνσης οικονομικής δραστηριότητα επίσης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με τα τελωνία. Η Κομισιόν θα αναθεωρήσει τον τελωνιακό καονισμό για τις ελεύθερες ζώνες. Μέχρι στιγμής ε, δεν ε, το κάναμε. Τα μεμονωμένα κράτη ελέγχουν και εφαρμόζουν τα μέτρα ελέγχουν και αποφασίζουν ποιες αρχές ελέγχουν ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλε οι δραστηριότητε ε, σέβονται την τελωνιακή νομοθεσία και την υπόλοιπη νομοθεσία πέραν τη τελωνιακή. Για να αξιολογήσουμε όμω την κατάσταση, οι υπηρεσίε μου έστειλαν ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη στις 26 Οκτωβρίου ε, αν υπάρχουν κάποιες δράσεις για να μετριάσουν τα προβλήματα. Τώρα, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προβλήματα στι ελεύθερε ζώνε, μπορούμε να παρέμβουμε. Όχι. Οι εθνικέ αρχέ πρέπει να εφαρμόσουν σωστά όλου του κανόνε και πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλε οι επιχειρηματικέ δραστηριότητε και οικονομικέ δραστηριότητε σέβονται αυτού του κανόνε. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικέ αρχέ μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση μη συμμόρφωση με του κανόνε. Διάφοροι ευρωβουλευτέ με ρωτήσατε για τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο, για τη δίκαιη φορολόγηση και αν ε, επεκτείνεται εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ε, διασυνδεδμένες αγορές και οι βασικοί κανόνες ε, ελευθέρου εμπορίου και δίκαιου εμπορίου πρέπει να γίνουν σεβαστές, το BEPS. Εμείς, ε, από την άλλη, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε πολύ πιο ενσωματωμένη και ολοκληρωμένοι μεταξύ μα πολύ περισσότερο από άλλε ζώνε. Και επομένω θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η φιλοδοξία μου ω επίτροπο είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ηγετικό ρόλο για να αποτρέψει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ε, υπάρχει ε, συνεργασία με παγκόσμιες σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ώστε όλοι να σέβονται τα ίδια διεθνή πρότυπα, πρότυπα που εμείς οι ίδιοι εφαρμόζουμε. Τώρα, ο κατάλογος είναι απόλυτη προτεραιότητα της, των φορολογικών αρμοδιοτήτων και θα ήθελα τρία πράγματα. Καταρχάς να εγκριθεί γρήγορα, δηλαδή τώρα, αρχές ε, Δεκεμβρίου, καμία καθυστέρηση δεν είναι αποδεκτή. Δεύτερον, να είναι αξιόπιστη, αξιόπιστος. Δεν θέλω να σας δώσω ένα νούμερο, δεν σας λέω ότι αν έχεις 12 χώρες ε, είναι αξιόπιστη και αν έχεις 8 ας πούμε δεν είναι αξιόπιστη. Φυσικά με, ένα, με μια χώρα δεν είναι αξιόπιστη. Ε, πάντως θέλουμε αξιόπιστο κατάλογο, που σημαίνει ότι όλες οι χώρες που δεν ε, συμμορφώνονται με τα κριτήριά μας πρέπει να μπουν στον κατάλογο. Τελεία. Και επιπλέον θα, θα πρέπει να έχουμε κυρώσεις. Δεν θα υπάρξουν πάρα αυτά κυρώσεις και δεν θα τις προσδιορίσουμε πάρα αυτά, αλλά συν το χρόνο. Αυτά για τη λίστα, για τον κατάλογο. Τώρα, τι πρόοδος έχει γίνει. Ουσιαστική θα έλεγα σημαντική. Από τις πληροφορίες που έχω από την ομάδα τελωνιακού, ε, κώδικα δυνατολογίας συγγνώμη, ε, μου γεννάται μία αισιοδοξία. Αυτή η ομάδα ε, είναι υπεύθυνη για τον κατάλογο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα κριτήρια και τις προτάσεις που τα υιοθετεί το Συμβούλιο, αλλά ο κώδικας δυνατολογίας κάνει την υπόλοιπη δουλειά για, την, για τον κατάλογο. Και τα πάει καλά. Τώρα είναι και η ώρα και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους ούτως ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, γι' αυτό ας περιμένουμε τις αρχές Δεκεμβρίου. για τον έλεγχο των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, που είναι ένα θέμα που μας ανισχύει πάρα πολύ. Καταρχάς, ε, καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών μας, χώρες που μερικές, ή των χωρών τέλος πάντων που μερικές φορές δεν μπορούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και να... Και επιπλέον ε, χρηματοδοτεί τρομοκρατία και άλλε εγκληματικέ δραστηριότητε η διακίνηση αυτή. Γι' αυτό ακριβώ πιστεύω ότι η πρόταση που υιοθετήθηκε στι 17 Ιουλίου θα σταματήσει την, το λαθρεμπόριο των πολιτιστικών αγαθών που εξάγονται παράνομα από τις χώρες τους ε, μέσω ενός ε, συστήματος ελέγχου των εισαγωγών. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις, δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες, απάντησα τις περισσότερες, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξουν ε, μαθήματα κατάρτισης για τελωνιακούς, τελωνιακούς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία και πρέπει να γίνει και μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση όλων εκείνων που πουλάνε και αγοράζουν ε, έργα τέχνης. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε την οικονομική αυτή δραστηριότητα, αλλά μόνο την παράνομη διακίνηση, το λαθρεμπόριο. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πλήξουμε το εμπόριο μοντέρνας τέχνης. Γι' αυτό μιλάμε για πολιτιστικά αγαθά που είναι τουλάχιστον 250 ε, χρόνων. Γιατί? Γιατί και η UNESCO λέει ακριβώς το ίδιο. Αυτή την ηλικία βάζει. Και γιατί αυτά τα πολιτιστικά αγαθά ακριβώ προσπαθούν να διακινήσει το, διακινήσει ISIS. Η πρόταση γενικά είναι ισορροπημένη. Περιμένουμε τη δική σα έκθεση βέβαια, την αξιολόγησή σα και τι προτάσει σα. Τώρα, αυτέ οι προτάσει πώ εντάσσονται ε, και συνδέονται με τις παγκόσμιες τάσεις. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλήσεις σε διεθνές επίπεδο για άμεση δράση κατά του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αγαθών, ειδικά όταν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η τρομοκρατία. Υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις όπως ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων, η UNESCO και διάφορα διεθνή βήματα όπως το G7 ας πούμε, που έχουν υιοθετήσει τάσεις και τις έχουμε συζητήσει. Η τάση είναι να ενισχύουμε τους ελέγχους κατά την εισαγωγή καθώς και την αποθήκευση στις ελεύθερες ζώνες. Ε, τώρα, ε, οι τελωνιακές αρχές ισχύζονται διότι είναι φιλικές προς τις α, επιχειρήσεις. Νομίζω ότι τα τελωνία πρέπει να βρουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο εμπόριο και στην διευκόλυνση του εμπορίου και την ε, διασφάλιση της ασφάλεια των αγαθών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν διάφορα μέσα για να το κάνουν αυτό. Καταρχά έχουν μόνιμες επαφέ με τους εμπόρους για τελωνιακά θέματα. Υπάρχει επίσης ε, ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας που έχουμε, είναι ένας ε, ορισμός που έχουμε εμείς ε, και έχει διευκολύνσει αυτός. Επίσης υπάρχουν οι τελωνιακές διασαφήσεις το 2015 91% των ε, εισαγωγικών ε, τελωνιακών διασαφήσεων διεκπεραιώνονταν μέσα σε, ένα, σε μία ώρα. Πάρα πολύ αποτελεσματική δουλειά. Τώρα, ποιες διευκολύνσεις έχουμε για το νόμιμο εμπόριο. Ε, υπάρχουν πολλές απλουστεύσεις ε, για το πώς θα υποβάλει κανείς τελωνιακή διασάφηση. Τις έχουμε εγκρίνει και θέλουμε να τις εφαρμόσουμε για την καλή φορολογική διακυβέρνηση στις εμπορικές ε, συμφωνίες. Σας απασχολεί όλους. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι δεν είμαι ο αρμόδιος επίτροπος για, το εμπόριο. Θα το πω στην ε, φίλη μου τη Σεσίλια Μάτσομ. Όλες οι ερωτήσεις σας σχετικές με το εμπόριο και τις παρατηρήσεις σας και, τους, και τις επικρίσεις. Αλλά η Κομισιόν συμφωνεί ότι χρειαζόμαστε καλή φορολογική διακυβέρνηση στι συμφωνίε μα με άλλε χώρε. Γι' αυτό στην εξωτερική στρατηγική θέλουμε να επικαιροποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη ρήτρα για τη φορολογική διακυβέρνηση στι διεθνεί συμφωνίε. Έχουμε τον κώδικα διοντολογία, ο οποίο επίση εργάζεται επί μια πιο ισχυρή ρήτρα και πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα φτάσουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Δεν αποφασίζουμε μόνο εμείς, το ξέρετε, παρότι ξέρουμε ότι έχουμε το μονοπόλιο διαπραγματεύση και διαπραγματευόμαστε εν ονόματι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξουν εμπορικέ ε, κυρώσει. Δεν τι έχει συζητήσει ο κώδικα διοντολογίας, ο του κώδικα διοντολογίας σε αυτή τη φάση. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, συζητήσει φορολογικά αντίμετρα. Ε, μπορούν να υπάρξουν και άλλα μέτρα, αλλά κατά την άποψή μου ε, το πιο σημαντικό πράγμα είναι τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για τα μέτρα. Τα, εμπορικά, τα μέτρα συναφή με το εμπόριο μπορεί να είναι ισχυρό εργαλείο ε, κατά των χωρών που παίζουν παράνομα, που δεν το παίζουν με βάση τους κανόνες. Το, βασικό είναι ότι τα αντίμετρα δεν θα πρέπει να ε, θέτουν να αμφιβόλω τις εμπορικές σχέσεις μας με τις ίδιες χώρες ή να έρθουν σε αντίθεση με την πολιτική μας, την εμπορική. Όταν κοιτάξετε τον κατάλογο μπορείτε να δείτε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Δεν θέλω όμως να προδικάσω οτιδήποτε και να μιλήσω για πράγματα που δεν ξέρω ή δεν μπορώ να φανταστώ η Κομισιόν θα δώσει, θα δημοσιοποιεί κάποιες φορολογικές πληροφορίες, τελωνιακές πληροφορίες. Ναι, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, ούτως ώστε να εντοπίζουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες εισάγουν αγαθά ή παράγουν αγαθά τα οποία δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα άκουσα τις προτάσεις σας. Η Ολομέλεια έχει ένα υιοθετήσει ένα ψήφισμα για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας που ζητάνε από την Κομισιόν να να δώσει πρόσβαση σε δεδομένα που συλλέγουν τα κράτη-μέλη, πρόσβαση δηλαδή στον κόσμο. Τα τελωνιακά όμως δεδομένα ε, υπόκειται στην προστασία με τον ίδιο τρόπο και τα προσωπικά δεδομένα, γιατί είναι ευαίσθητε πληροφορίε. Επίση, η πρόσβαση στα θελωνιακά δεδομένα, όπω οποιασδήποτε πληροφορίε που έχουν οι δημόσιε αρχέ των κρατών μελών, είναι θέμα εσωτερική ένωμη τάξη, εθνική ένωμη τάξη. Και η Κομισιόν νομίζει ότι ο καλύτερο τρόπο για να δράσουμε είναι να συνδέσουμε ή μάλλον να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα μέσω τη εθνική νομοθεσία του. Τι θα κάνουμε ούτως ώστε οι online πλατφόρμες να πληρώνουν ε, του φόρου όταν λειτουργούν, φόρους που του αναλογούν. Η οικονομία στο μέλλον θα είναι όλο και πιο ψηφιακή και θα πρέπει να προσαρμόσουμε το φορολογικό μα σύστημα για να το λάβουμε υπόψη μα αυτό. Η βέλτιστη λύση θα ήταν ε, μια παγκόσμια λύση. Όμω εμεί ε, θέτουμε αυτό το θέμα στο πλαίσιο του ΩΣΑ, ακριβώ γι' αυτό. Πρέπει όμω να βρούμε και λύσεις για την εσωτερική αγορά. Ειλικρινά σα λέω ότι για μένα η καλύτερη λύση είναι ε, η CCCTB, η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση ε, για των εταιριών. Μπορούμε να κάνουμε όμως και πιο συγκεκριμένες προτάσεις, γι' αυτό θα δούμε όλες τις επιλογές και θα ετοιμάσουμε μια πρόταση ή μια σειρά από προτάσεις την άνοιξη του 2018. μετά την ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε το Σεπτέμβριο του 2017, που δίνει κάποια στοιχεία για αυτό το θέμα. Ε, μου με ρωτήσατε για την αρμόνιση των φόρων από, άνθρωπου, από ανθρώπους που δεν είναι και φεντεραλιστές, ε, άκουσα αυτή την ερώτηση. Αν θέλετε να εναρμονίσετε τον ε, φόρο, θα πρέπει να αλλάξετε τους κανόνες του παιχνιδιού προς περισσότερη ολοκλήρωση, αν όχι προς ε, ομοσπονδία. Γιατί μας, τι μας μπλοκάρει σήμερα τα φορολογικά που φασίζονται με ομοφωνία. Άρα με ένα βέτο ο ένας σταματάει τη θέληση όλων. Αν θέλουμε λοιπόν ε, μια εναρμόνιση και μια Ευρώπη πιο φιλόδοξη, πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού και να πάμε από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ που το προτείνατε. Είμαι υπέρ τέτοιων ε, προβληματισμών. Και αυτή είναι και η απάντησή μου. Επιτέλους συμφωνούμε κιόλα. Ευχαριστώ για τη φεντεραλιστική σας πρόταση, που είναι πραγματικά κάτι πολύ προσφυλές σε Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επίσης ε, θα πρέπει να έχει μία ε, ενιαία εφαρμογή των δασμολογικών ζητημάτων. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η Κομισιόν θεωρεί πως σε κάποιες πρακτικές δεν συμφωνούν με την νομοθεσία της. Άρα υπάρχουν οι διαδικασίες κατά παραβάση, επί που ξεκινούν να κινούν για τέτοια κράτη-μέλη. Πάμε τώρα στη μακροοικονομική βοήθεια. Καταρχάς για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ε, βοήθεια αυτή, για την Ουκρανία και την Ινδονησία είναι θετική. Γενικά το πακέτο, όπως ξέρετε αυτοί ε, οι εκθέσεις δημοσιεύονται με την απάντηση της Κομισιόν σε κάθε παρατήρηση του συνεδρίου. Θα πρέπει να δείτε ότι σε δύο σημεία υπήρχε ένα θέμα στην Ουκρανία με εξέπληξε που ήταν κάπως αυστηρή για τη δεύτερη εκταμίευση του προγράμματος. Αυτό δεν είχε αναλυθεί ε, στην έκθεση ε, ως προς το διάστημα 31 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 μετά φτάσαμε μέχρι τον Απρίλιο του 2017 από εκεί και πέρα να πω ότι η Κομισιόν πάντοτε είναι διαφανής και συγκεκριμένη στη δουλειά της ε, Τώρα, για την άλλη χώρα, νομίζω είναι πολύ αργές ε, οι διαδικασίες στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο όχι στην Κομισιόν. Έτσι λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο μας ζητά να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Ε, πραγματικά συμφωνώ πλήρως με το να γίνει μια τέτοια συζήτηση μαζί σας. Για την Ουκρανία Το θέμα αυτής της εκταμίευσης δεν είναι εύκολο. Η διαθεσιμότητα της μακροοικονομικής βοήθειας ε, λίγη στα τέλη του έτους. Ε, σύντομη λοιπόν προθεσμία. Και παραμένουν κάποιοι όροι που δεν πληρούνται πλήρως για αυτήν την εκταμείευση. Το συναντήσαμε, συναντήθηκα ήδη με τον Υπουργό. Σήμερα το απόγευμα θα ξανασυναντηθούμε και θα τα πούμε για άλλη μία φορά. Εφόσον έχω ακούσει και τους στόχους της δικής σας επιτροπής και άλλων, να πω ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον θα κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσουμε στη σωστή κατεύθυνση, αφού είναι κοινή στόχη, όμως ε, πρέπει να έχουμε και μια ισορροπία και η αιρεσιμότητα να τηρείται και η Ουκρανία να βοηθηθεί. Κάποιοι με ρωτήσατε για το πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για την εφαρμογή των ε, όρων στην Ουκρανία και σε άλλες ε, τέτοιες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες. Σίγουρα, συμφωνώ μαζί σας, ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στη γειτονία μας οι χώρες εταίροι εφαρμόζουν τους όρους, γιατί καταρχάς είναι σημαντικό και βασικό για τις ίδιες τις χώρες. Δεν θέλουμε να δημορίσουμε τον κόσμο, απλώς θέλουμε να τον βοηθήσουμε να προοδεύσει ως προς την οικονομική σταθερότητα, γιατί η δημιουργία θέσεων εργασίας υφίσταται μόνο όταν υπάρχουν και άλλες διαδικασίες ήδη που λειτουργούν. Ε, μία από αυτές είναι η μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση όμως πρέπει να γίνεται από την ίδια τη χώρα, να είναι η χώρα ο ιδιοκτήτης των αλλαγών των μεταρρυθμίσεων και ο εμπνευστή. Για, τις εμπορικές, ε, για τους εμπορικούς δεσμούς, ε, ένας τε, η βοήθεια αυτή είναι ένας τέτοιος δεσμός, αλλά είναι κυρίως ένα εργαλείο οικονομικής σταθεροποίησης. Αυτό είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Θα συζητήσουμε με τη Σεσίλια Μάστρομ λοιπόν με το ίδιο πνεύμα που συζητήσαμε και τα προηγούμενα, αλλά μάλλον πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτική για τη Μολδαβία τώρα. Παρόλο που υπάρχει ε, σημαντικό κομμάτι δουλειάς που πρέπει να γίνει ακόμα, αναγνωρίζω εδώ ότι η Μολδαβία έχει κάνει πρόεδρο σε μία σειρά κρίσιμης σημασίας μεταρρυθμίσεων. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα πάταξη της διαφθοράς. Έχουν εγκρίνει την Εθνική Στρατηγική για την Ακαιρότητα και την πάταξη της διαφθοράς. Όμως, η Κομισιόν, σε συνεργασία με τις αρχές, μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας, της βοήθειας αυτής, θα προσπαθήσει να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Μολδαβία, ώστε να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό της μεταρρυθμίσης για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας που διασφαλίζουν όχι μόνο τη μεταρρύθμιση αλλά και την εφαρμογή. Θα συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό ε, της Μολδαβίας σήμερα. Είναι η μέρα μου σήμερα για την μακροοικονομική βοήθεια, οπότε θα προσπαθήσω να πετύχω πρόοδους και σε αυτό το θέμα. Για το Brexit δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που ήδη γνωρίζετε. Ο κύριος Μπαρνιέ είναι ο βασικός διαπραγματευτής, μάλλον ο μόνος που μιλά στην Κομισιόν για αυτό το θέμα. Δεν θα δώσω λεπτομέρειες, απλώς να πω ότι πιστεύουμε στεναρά πως πρώτα πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι, ο οικονομικός διακανονισμός, ε, τα δικαιώματα των πολιτών και το θέμα των συνόρων με την Ιρλανδία και μετά μπορούμε να περάσουμε σε συζήτηση για τις μελλοντικέ μας σχέσεις και τη σχέση που θα έχουμε. Τέλος, τρία πιο γενικά ερωτήματα που θέλω να απαντήσω πολύ γρήγορα για το FTT. Δεν είναι μυστικό που ότι είμαστε υπέρ. Υπήρξε πρόταση από την Κομισιόν, δεν υπήρξε συμφωνία. Και έτσι τώρα έχουμε την ενισχυμένη συνεργασία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στις 15 Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου έγινε μια συζήτηση, ανάλυση των επιπτώσεων του, exit, του Brexit σε αυτή τη ε, διαδικασία και είπαμε να γίνει λίγο πιο αργή η διαδικασία. Τα 10 κράτη-μέλη τα οποία μπλέκονται έχουν ε, φτάσει σε συμφωνία για το βασικό στοιχείο, ποια είναι η κοινή οντότητα. Ε, αν θέλουν μια ευθυτή μπορούν να την έχουν άμεσα. Είναι στο δικό τους ε, γήπεδο το μπαλάκι κατά τη γνώμη μου. Είτε σταματούν είτε γίνεται η συμφωνία. Και δύο τελικές ερωτήσεις, τελευταίες ερωτήσεις. για την συνταλλαγματική ισοτιμία. Συμφωνώ με τον κύριο Μορέλ, με κάθε σεβασμό που έχω στο κοινοβούλιο. Δεν πρέπει απλώς να απλουστεύουμε τα πράγματα. Γιατί δεν μας δείχνει τίποτα ότι η ισοτιμία του ευρώ σήμερα θα είναι φραγμός στο εμπόριο. Ξέρετε ποια ήταν η ισοτιμία στο παρελθόν. Έχουμε παρατηρήσει επίσης ε, ότι δεν υπάρχει κάποια μείωση της παραγωγής, ότι υπάρχει μια ε, ανταγωνιστικότητα ανευπροηγουμένου και δεν έχουμε πρόβλημα στην βιομηχανία λόγω του ευρώ. Δεύτερον, το πραγματικό πρόβλημα για να το θέσω σωστά, είναι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Ντομπρόφσκης, ε, ο συνάδελφός μου, παρουσίασε την άποψη της Κομισιόν, αλλά και τον μηχανισμό επαγρύπνησης που έχουμε για αυτές τις ανισορροπίες. Υπάρχουν οι ελληματικές χώρες, έχουν έλλειμμα στο προϋπολογισμό τους είτε στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών, συναλλαγών μάλλον, ε, όμως υπάρχουν και άλλα ελλείμματα. Χώρες που έχουν ε, ένα τρέχον πλεόνασμα ε, που θα μπορούσε να βοηθήσει για την ευημερία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της μέσα από περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές. Δεν αναφέρομαι σε κανέναν προσωπικά, αλλά εντάξει, η Γερμανία και η Ολλανδία συνήθως αναφέρονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές οι ανισορροπίες είναι αμοιβέ. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για κάτι άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας ε, για να έχουμε έναν πιο συγκεκριμένο και στοχευμένο διάλογο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ακρόαση. Να πω για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι αυτή η διεθνής ατζέντα για μένα. Είναι δική μου. Και είμαι διαθέσιμος να έρθω εδώ όποτε με ε, ζητήσετε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Και έχω και ένα αίτημα. Να εγκριθεί γρήγορα η πρόταση για το εμπόριο πολιτιστικών προϊόντων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε πολύ και καλή τύχη στις συνομιλίες που θα έχετε με τον Υπουργό, όπως μας είπατε. Για τα υπόλοιπα θα παραμείνουμε σε επαφή. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 19 τώρα τη ημερήσια διάταξη. Διάφορα. Έχετε διάφορα. Παρακαλώ, κύριε Ντάρθμορτ. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω, παρακαλώ. Συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύσατε αυτή την ε, τελευταία συζήτηση. Γιατί έτσι είχαμε χρόνο, επαρκή χρόνο, να θέσουμε τις ερωτήσεις μας, τα σχόλιά μας κλπ. Όμως χτες, στην ευρύτερη συζήτηση που είχαμε με τόσους διακεκριμένους, έκανα μια πολύ σύντομη παρέμβαση, 45 δευτερόλεπτα, αλλά θα ήταν προτιμότερο, θα ήταν καλό αν οι συνάδελφοι είχαν περισσότερο χρόνο να συμμετάσχουν σε αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις με το διακεκριμένο πάνελ. Ίσως σε μια συνάντηση συντανιστών θα έπρεπε να τεθεί αυτό. Έτσι, οι σκέψεις είναι αυτές που λέω για προβληματισμό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα τα συζητήσουμε εδώ οι δυο μας και θα επανέλθουμε. Ωραία. Σημείο 20. Προσεχή συνεδρία 28 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.